Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στο τελευταίο τμήμα της ε, συνεδρίας της ε, Επιτροπής μας. Όσοι ήταν στο, στην μαραθώνια συνεδρία σήμερα το πρωί, ελπίζω να ενδυναμώθηκαν μεταξύ, να είναι έτοιμοι για ένα πολύ σημαντικό φάκελο. την πρόταση οδηγίες για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο Χάιντ Φλόρεντ είναι ο εισηγητή μα, εργάστηκε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν συμβαστικέ προτάσεις και μπορούμε αμέσω να περάσουμε στην ε, συμβαστική τροπολογία παριθμών 1. Ποιο είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σωματοποιημένη, παγιωμένη πρόταση υπερθμών 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παλιωμένη τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε συμβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά, με μονομένες τροπολογίες. 58 Βίλς. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εξήντα. Τον τώρα Παναγιώτοφ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Διαδικαστικό. Δεν ξεχάσατε να ε, ε, δεν ξεχάσατε να υποβάλλετε ψηφοφορία και την 59. Ναι, ε, δυστυχώς κατέπεσε γιατί εγκρίναμε την 58. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Μετά, καταπίπτουν πολλές από τις τροπολογίες, γιατί εγκρίναμε τις συμβαστικές και έχουμε άρθρο 2 παράγραφο 4 10 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Εβδομήντα πέντε, ο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εβδομήντα έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ ε, τα φτάσουμε την 80 79-80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε. Την 81. Ηλεκτρονικός ελέγχος για την 81. Δύο σοσιαλιστές υπάρχουν. Ένα ένας Ακόμα ένα, εντάξει τώρα. Λοιπόν, 33 υπέρ, 23 κατά. Εγκρίθηκε. 84 υπέρ. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 αποσύρθη 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άπλες απεσύρθη. 12 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 96 και 97. Ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 98 και 99 και 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 101 και 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται επίσης. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εκατόν οκτώ αριστερός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. δεκαοκτώ υπέρ κατά απεχές να ελέγξουμε για την 118 πέρας πληροφορίες υπέρ εγκρίνεται λοιπόν περνάμε. Άρθρο 6 παράγραφος 1, 125, Παναγιώτοφ, υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Άρθρο 7, παράγραφος 1α, Σνέλχαρτ, 140. Υπέρ τη 140. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. Άρθρο 8, παράγραφος 2α. Σαμπίνα Βίλς, τροπολογία 165, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 167 του εισηγητή, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 του εισηγητή, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 170. Χριστέβη, υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 171, υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. 21, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 172 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 187 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται Εκατόν ογδόντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε, να ελέγξουμε την 192 Άνς από την SD και άν από το ΕΤΣΕΡ ε, υπεράριθμη. Τώρα είμαστε εντάξει. Ενεκρίθη 31 προς 27. Εκατόν τρία, υπέρ. Κατά. εποχέ.

αποχές έλεγχος 194 ελέγχουμε πέρας απερίφθη 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 201. 201. Υπέρ. 201 σκυλακάκες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 204. Χριστέφης υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 205. Λεπάζ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 211 και 207. Davis και τελάνε. υπερ Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 211-207. Έλεγχος. Ένα από το υπεράριθμο. Ωραία. Πέρα. 35 προς 25. Εγκρίνεται. 210. Βάσκερ Βεκράμε, Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Mm -hmm. 218 γκροστέτ σουλή, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 219 Γκέρλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 220 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 222-242 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 223 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 224. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 230 και 240 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 231 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 232. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 234. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 233. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 235 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 236, 237, 238, 239 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 241 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 243. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 244. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 245 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 246 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 247 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 248 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και αυτή. Alle Davies sind angenommen. Also, wir machen weiter. 200 Λοιπόν, συνεχίζουμε. 250 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 249 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 251 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται επίσης ε, τώρα. 253. Τρεμόπουλος υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 254. Σφιέλνα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 255. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται επίση. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 256 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 257 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 258 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 259 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 260 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 261 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επίσης ολόκληρη σειρά ενεκρίθη δεν βλέπω αν από την Ελλάδα. Καλά. 40 äh, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 263 και 41 κατά τμήματα, το πρώτο τμήμα. Λοιπόν, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 263 δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. εποχές, Απορρίπτεται. 263 τρίτο τμήμα. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Εποχές βέβαια ρώτησα. 41 δεύτερο τμήμα, υπέρ. Α, έχει κατα... καταπέσει. Καλώς. Ναι, ναι. Και φτάνουμε στις ειδουλικές σκέψεις. Τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 50 50 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά ε, εγκρίνεται 56 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται και 57 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Α, γλίγορα τελειώσαμε. Πολύ ωραία. Θαυμάσια. Τώρα τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά για το σύνολο της έκθεσης. Άρχη ψηφοφορία. S και J ένας υπεράριθμος. Εντάξει τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. 54 υπέρ, μία ψήφος κατά και τρεις αποχές. Και η δεύτερη ψηφοφορία, το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, πάλι ηλεκτρονικά, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίες. 51 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά και τρεις αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή Καλχάης Λόρενς. Και συγχαρητήρια και σε όλους τους οικειώδεις που συνεργάστηκαν και στη γραμματεία που τα προετοίμασαν τα πράγματα τόσο ωραία. Και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της της διάταξης. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Und zwar die Debatte über Deepwater Horizon. Τη συζήτηση για το Deepwater Horizon και την πατρελοκυλίδα στον κόλπο του Μεξικού. Deepwater Horizon Λοιπόν, Deepwater Horizon και πετρελαιοκυλίδα στον κόλπο του Μεξικού. All electronic waste people who like to continue the votes and the debate out. Ε, εκείνοι που ενδιαφέρονται για τα ηλεκτρονικά και τα, ηλεκτρο... και τα ηλεκτρικά απόβλητα να συνεχίσουν συζητήσεις του παρακαλώ εκτός της αιθούσης. okay? Yes, yes. Wonderful. PPE, are you clear? So. Λοιπόν, αν είμαστε όλοι έτοιμοι, θα δώσω το λόγο στον Νίχια Τζίβερ. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Auch von meiner Seite noch δεν ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή για το πολύ καλό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ε, από την άλλη μεριά έχουμε ένα πολύ επίγον περιβατολογικό πρόβλημα, όχι ενώπιον των θύρων ίσως, αλλά πολύ σημαντικό για όλο το ατλαντικό περιβάλλον. Όλα αυτά, όπως ξέρετε, από διάφορες εικόνες που βλέπουμε στην τηλεόραση, λαμβάνει χώρα στον κόλπο του Μεξικού και θα πρέπει να κάνουμε νομίζω καταρχήν μια συζήτηση εδώ για το θέμα της εξόριξης πετρελαίου σε ακραίες περιπτώσεις. Εδώ είχαμε μια πλατφόρμα εξόριξης στη θάλασσα που εξεράγει, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε γενικά την εξόριξη πρώτων υλών για την ενέργεια κάτω από πολύ επικίνδυνες ε, προϋποθέσεις και θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το νομικό πλαίσιο που χρειάζεται όσον αφορά ιδίως την ασφάλεια και τι θα πρέπει να κάνει σχετικά ο νομοθέτης. Εγώ πολλά βέβαια έχω μάθει από τα ΜΜΕ. Από όσο ξέρω, οι νομοθετικέ διατάξει τη ΕΠΑ δεν είναι τόσο αυστηρέ όσο εδώ στην Ευρώπη, αλλά αυτό ήταν ενδιαφέρον να μα πει η Κομισιόν πώ εκτιμάει εκείνη την κατάσταση και πού θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση στην Ευρώπη. Ένα άλλο θέμα είναι ένα ταμείο που θα μπορούσε ίσως να καλύψει τις ε, ζημιές. Η εταιρεία πετρελοδών BP υποσχέθηκε ότι θα δημιουργήσει ένα τέτοιο ταμείο. Θα πρέπει όμως κάτι να κάνουμε για να μην εξαρτώμαστε από την καλή θέληση κάποιες εταιρείες στο μέλλον γιατί νομίζω ότι το πλήγμα στο περιβάλλον είναι πολύ πιο σκληρό από ό,τι ακούμε. Συνήθως ε, συζητάνε μόνο για το πλήγμα στη βιομηχανία. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τι θα γίνει αν συνεχίζει να εχύνεται το πετρέλαιο. Θα μπορούσε η Ευρώπη ίσως να πληγεί μέσω των ρευμάτων του ρεύματος του κόλπου Μεξικού Φερρυπίν. Και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Εμείς σε Επιτροπή ΕΝΒΗ θα πρέπει νομίζω να δημιουργήσουμε μια άποψη και ενδεχομένως να προετοιμάσουμε και ένα ψήφισμα για την επόμενη σύνοδο ολομελίας, μια που το θέμα είναι τόσο τόσο σημαντικό και αφορά όλο το τομέα της, ε, των πρώτων υλών ενέργειας. Και θα μπορούσαμε έτσι να συμβάλλουμε σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ρίχια Τσέβερ, λέει Πρόεδρος. Υπάρχει μια σειρά ερωτήσεων προς την Κομισιόν. Θα πρότεινα λοιπόν ο κύριος Γιάννεχ της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργεια να απαντήσει σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Παρακαλώ, αν θέλετε να τοποθετείτε από αυτόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιβάλλοντος διότι συμπεριέλαβε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξή της. Να υπενθυμίσω την παρουσία του Επιτρόπου στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Πριν από ένα μήνα σας ε, είπε τι δράση ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από την καταστροφή στον κόρπο του Μεξικού και εκεί κάλεσε και το Κοινοβούλιο να συνεργαστεί στενά με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα επόμενα βήματα. Επομένως, εκτιμούμε ιδιαίτερο την πρωτοβουλία της Επιτροπής σας. Ε, μας χαροποιεί το γεγονός ότι μπορούμε να ανταλλάξουμε ε, απόψεις και προσβλέπουμε και σε διάλογο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε πρακτικά συμπεράσματα. Θα πρέπει να πω, βέβαια δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το υπενθυμίσω, αλλά θα πρέπει να πω ότι συμπονούμε τους πληγέντες ε, της καταστροφής του Μεξικού ε, και του κόλπου του Μεξικού και φυσικά και σε επαγγελματικό αλλά και προσωπικό επίπεδο ε, νιώθουμε ε, θλίψη για τα όσα συνέβησαν. Αυτά εισαγωγικώς. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίσουμε το θέμα είναι να σας παρουσιάσω μία εικόνα των δράσεων που έχει αναλάβει μέχρι τούδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτά τα οποία είναι εν εξελίξη και εσωτερικό στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και εξωτερικό σε σχέσεις με άλλα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και με άλλους ενδιαφερομένους και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν ε, σας αναφέρω επιγραμματικά τις δράσεις αυτές, να κάνω ένα-δυο σχόλια για την κατάσταση στον κόλπο του Μεξικού Πρώτον, γνωρίζουμε ότι η καταστροφή είναι ακόμα ανεξελίξη. Η έρευνα η οποία ξεκίνησε από τις Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά νομίζω και όλες οι υπόλοιπες αναλύσεις είναι ακόμα και αυτές εν εξελίξη και νομίζω ότι τα τελικά αίτια της καταστροφής δεν έχουν καθοριστεί, δεν υπάρχει ένα τελικό απόρισμα και αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. όταν εξετάσουμε ποιε θα είναι οι κατάλληλε δράσει ω ανταπόκριση σε αυτή την καταστροφή. Δεύτερον, θα πρέπει να σκεφτούμε και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων που διεξάγονται στον κόλπο του Μεξικού και στα αντίστοιχα φαινόμενα στην Ευρώπη. Ο κλάδος μας έχει δώσει στατιστικά στοιχεία, λέμε ότι το βάθος στο οποίο γίνονται οι αντίστοιχες έρευνες στην Ευρώπη είναι πολύ μικρότερο από το βάθος που είχαμε στην πλατφόρμα Deepwater Horizon. Από τις πληροφορίες που έχουμε από τον κλάδο, τις οποίες επαληθεύουμε αυτή τη στιγμή με τις εθνικές αρχές ε, των κρατών μελών αλλά και με άλλα κράτη-μέλη, και εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση ο κλάδο ε, συνήθω δραστηριοποιείται σε βάθο 100-200 ε, μέτρα, ενώ ε, έχουμε κάποιε επιχειρήσει σε βαθύτερα νερά, αλλά νομίζω ότι η βαθύτερη είναι η περίπου 700 μέτρα, που είναι περίπου τα μισά από όσα έχουμε στο Deepwater Horizon. Έχουμε λοιπόν μία σαφή ένδειξη από τον κλάδο και αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε Ορισμένες φορές οι συνθήκες ε, εντός των πηγών μπορούν να συγκριθούν με τα όσα γίνονται στον κόλπο του Μεξικού. Δηλαδή φαίνεται ότι γίνονται γεωτρήσεις όλο και βαθύτερα και όσο βαθύτερα γίνονται οι γεωτρήσεις τόσο μεγαλύτερες πιέσεις αντιμετωπίζονται. αλλά συνήθως ε, έχουμε επιχειρήσεις σε βάθη τα οποία συνήθως μπορούν να φτάσει ο άνθρωπος και σημαίνει ότι είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο αποδετικοί ως προς τη διαχείριση ε, μιας κρίσιμης κατάστασης που μπορεί να προκύψει εκεί επί τόπου σε σχέση με αυτά που θα βλέπουμε καθημερινά στη τηλεόραση να συμβαίνουν στον κόλπο του Μεξικού όπου έχουμε χειρισμό μηχανομάτων με τηλεκίνηση και υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι περιορισμοί από πλευράς πίεσης ε, σε αυτό το βάθος Λαμβάνοντα κλπ. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τις συνθήκε που επικρατούν, ε, εμείς ε, αναλάβαμε δράση πάρα πολύ γρήγορα μετά από τη διαπίστωση της καταστροφής. Ε, αρχίσαμε να έχουμε κάποιες εσωτερικές διαδικασίες, ε, ε, ε, αναθεώρηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Αυτά τα είπα και στην εισαγωγή μου υπάρχει ένα πλήρες φάσμα ευρωπαϊκής νομοθεσίας που ισχύει για τις γεωτρήσει και από παράκτιες ε, ε, πηγές. Ε, αυτά όλα συμπληρώνονται με εθνική νομοθεσία και με νομοθεσία που αφορά τεχνικά θέματα, θέματα ασφάλειας, λειτουργική ασφάλειας, προστασία προσωπικού, καθώς επίσης και προστασία του περιβάλλοντος και προστασία από πετρολοκυλίδες ή ζημίες, καθώς επίσης και θέματα αποζημιώσεων και ευθυνών ε, για να μπορέσουμε να αποδώσουμε ευθύνε σε περίπτωση που έχουμε ένα καταστροφικό ε, γεγονός, καθώς επίσης και το ποιος έχει την ευθύνη για καθορισμό και ε, απορρίπανση στη συνέχεια. Όλα αυτά είναι πλήρη και καλύπτουν ε, ε, καταλήλως όλα όσα μας αφορούν. Ε, ξεκινούμε και μια εσωτερική αναθεώρηση με τις διάφορες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τα διάφορα τμήματα του κεκτημένου και γίνεται ένας έλεγχος για να δούμε τι υπάρχει και πόσο καλά λειτουργεί. Ξεκινά και η σύσταση μιας ενδουπηρεσιακής ομάδας, αφού κάνουμε αυτή τη διαδικασία που σας ανέπτυξα, θα κάνουμε και αυτή την ομάδα, θα συσταθεί αυτή η ομάδα για να υπάρχει συντονισμός, ίσως και σε νομοθετικό πλαίσιο, λαμβάνοντα υπόψη βέβαια και το γεγονό ότι οι έρευνε είναι εν εξελίξη, επομένως ε, εάν υπάρχουν αδυναμίε ε, στην νομοθεσία θα τι ε, διαπιστώσουμε, θα δούμε κατά πόσον είναι οι κατάλληλε. και εάν θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να προληφθούν τα αίτια τα οποία προκάλεσαν το ατύχημα, θα ληφθούν και αυτά τα μέτρα. Έχουμε και μηχανούς, ε, μηχανισμούς ανταπόκρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά όλα βέβαια όπως σας είπα συμπληρώνονται πάντα και με τα μέτρα που έχουμε σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν ανάλογα εργαλεία και σε εθνικό επίπεδο κυρίως από, από χώρες που έχουν ε, επιχειρήσεις γεωτρήσεων αλλά ε, θεωρούμε ότι αυτά μπορούν να προσδώσουν επιπλέον αξία στην ευρωπαϊκή νομοθεσία εάν μας ενδιαφέρει κάτι παραπάνω. Υπάρχει και ένας ειδικό οργανισμός ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Ναυτιλιακής Ασφάλειας, της ΕΦΣΑ. Έχουμε και συναδέλφους από την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση εδώ. Πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος ε, έχει πολλά μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση των πετρελοκυλίδων και ε, να βοηθήσουν χώρες που αντιμετωπίζουν καταστροφές, καθώς επίσης ε, και συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση πολιτικής προστασίας που είναι και αυτοί αρμόδιοι και θα μπορέσουν να ε, συντονίσουν τις δράσεις τους με τις δικές μας. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε έναν έλεγχο της νομοθεσίας, της εσωτερικής μας νομοθεσίας για να δούμε αν έχουμε όλα όσα μας χρειάζονται αλλά ξέρουμε ότι οποιοδήποτε ρυθμό, ε, ρυθμιστικό καθεστώ και να έχουμε, ακόμα και στο μέλλον, δεν θα μπορέσει να μα δώσει 100% ε, διασφαλίσει ότι όλα λειτουργούν καλά. Ένα σύστημα είναι καλό εάν συμμορφούνται όλοι προ του κανόνε του. Οποιαδήποτε προσέγγιση λοιπόν ακολουθήσει ο κλάδο ή οποιοδήποτε, οποιοδήποτε από του ενδιαφερομένου θα πρέπει να συμμορφείται προ του κανόνε και θέλουμε ε, οι αρμόδιοι, οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο διάλογο. Ο Επίτροπος ε, ήρθε στην Ολομέλεια μαζί με την Επίτροπο Γεωργίευα συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του κλάδου που δραστηριοποιούνται στον τομέα στις 11 Μαΐου και τους έθεσαν κάποιες ερωτήσεις, κάποιες προφορικώς, κάποιες τους δόθηκαν γραπτός για να τις πάρουν μαζί τους για το σπίτι. Όλα αυτά γίνονται για να διασφαλίσουμε ότι ο κλάδος λαμβάνει όλα τα μέτρα διασφάλισης ώστε να προληφθούν κίνδυνοι για τους κινδύνους ε, στους οποίους θα μπορούσαν να εκτεθούν οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης από περιβαλλοντικής πλευράς. τον Ιούλιο προβλέπεται μια συνεδρίαση για να αναθεωρήσουμε τις απαντήσεις που θα λάβουμε από τις γραπτές ερωτήσεις που τους δόθηκαν. Ε, προβλεπόταν αρχικώς να συναντηθούν μετά από τρεις μήνες με τον κλάδο, αλλά επειδή η κατάσταση εξελίσσεται τελείως διαφορετικά, ε, μάλλον θα γίνει συντομότερη προθεσμία, γι' αυτό η συνεδρίαση θα γίνει μετά από δύο μήνες και εκεί Φυσικά θα γίνουν περαιτέρω συζητήσεις ε, για να μπορέσουμε να έχουμε ε, σαφείς επιπλέον πληροφορίες για το κατά πόσον δεσμεύονται ως προς την ασφάλεια. Μιλούμε επίσης με τους εθνικούς ρυθμιστές. Η πρώτη συνεδρίαση θα γίνει την Παρασκευή αυτή την εβδομάδα και στη συνέχεια μετά από κάποιες εβδομάδες θα έχουμε μια συνεδρίαση των ε, επικεφαλής ε, των ρυθμιστικών ε, ομάδων για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι ρυθμιστικές αρχές και οι εθνικές διοικήσεις επί των θεμάτων αυτών και τι απαραίτητες βελτιώσεις πρέπει να γίνουν ανάλογα με τα όσα θα προκύψουν από τους ρυθμιστικούς φορείς και το κατά πόσον θεωρούν ότι πρέπει να βελτιώσουμε το επίπεδο της ε, ασφάλειας και να ε, βελτιώσουμε και το επίπεδο των ελέγχων συμμόρφωσης από πλευράς ρυθμιστικών φορέων. Επίσης ε, και με εξωτερικούς ενδιαφερομένους εξετάζουμε τα θέματα της ε, παράκτιας ασφάλειας. Ε, το θέμα της ασφάλειας των παράκτιων γεωτρήσεων δεν ήταν βέβαια κάτι το οποίο αποτελούσε προτεραιότητα στο παρελθόν. Πολλές φορές είδαμε αρνητικές επιπτώσεις από άλλα σημεία της αλυσίδας του αργού πετρελαίου και των παραγωγών πετρελαίου σε θέματα διακίνησης, μεταφοράς κλπ. Το θέμα λοιπόν του κινδύνου για τις παράκτητες δραστηριότητε είναι ναι μεν καινούριο αλλά θέλουμε να το συμπεριλάβουμε στις συζητήσεις αλλά και στην Ευρώπη ε, υπάρχει το λεγόμενο Berlin Forum που είναι μια πλατφόρμα ε, την οποία χειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και θέλει να συγκεράσει ενδιαφερομένους στον τομέα και να μπορέσουν να συζητήσουν τα θέματα αυτά και εκεί θα τεθεί το θέμα της παράκτης ασφάλειας ως ε, προτεραιότητα και φυσικά θα το βάλουμε και στις ε, ε, συζητήσεις μας με τρίτους εταίρους, χώρες για παράδειγμα όπως οι ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Ρωσία και μπαίνει και στην ημερήσια διάταξη των πελημερών συζητήσεων με τις ε, χώρες του ΟΠΕΚ. Υπάρχει και μία υπουργική διάσκεψη τη Δευτέρα. Αυτό έχει μπει στην ημερήσια διάταξη λοιπόν ως ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουν. Υπάρχει και η ομάδα των χωρών ε, της συνεργασίας του κόλπου και θέλουμε να το συζητήσουμε και με αυτούς και από ό,τι ξέρουμε και το G20 θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Και θέλουμε λοιπόν να συζητήσουμε ε, στην πλατφόρμα αυτή και με τις χώρες του G20 για το θέμα της παράκτησης ασφάλειας. Αυτά λοιπόν εν είδη σύντομη σύνοψη. Βλέπετε τι κάνουμε και ως προς τις νομοθετικές μας δράσεις για να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε την καλύτερη δυνατή νομοθετική κάλυψη αλλά και ως προς μη νομοθετικές ε, διαδικασίες. Φυσικά θα ρωτήσετε αν υπάρχει κάποια απευθείας νομοθετική δράση η οποία αναλήφθηκε από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, Να σας πω και πάλι ότι πριν γνωρίζουμε ακριβώς τα αίτια της καταστροφής δεν θα γνωρίζουμε τι ακριβώς δράση πρέπει να αναλάβουμε για να έχουμε νέα πρότυπα και προδιαγραφές. Αλλά ε, ήδη έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ίσως μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι σαφές ή χρειάζεται τροποποίηση για να ε, ισχύει και για την ε, παράκτη ασφάλεια. Αν τυχόν καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα θα αναλάβουμε και τις ανάλογες δράσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, Κύριε Πανέκ, μιλήσατε εξ ονόματος της ΕΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ενέργειας. Ο κύριος Αρσένης είναι ο πρώτος ομιλητής στη συζήτησή μας. Παρακαλώ και μετά η κυρία Λεπάζ. Ε, Φαίνεται ότι δεν έχει τέλος ε, αυτή η καταστροφή. Κατασκευάστηκε η εξέδρα το 2001 παρόλα αυτά, δηλαδή είναι νέα η τεχνολογία, είναι πρόσφατη η εξέδρα. Ε, στα αμερικανικά η ύδατα δεν ξέρω πόσες εξέδρες ε, έχουμε, μήπως έχει τα στοιχεία Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γύρω στις 400 πρέπει να είναι. Ε, το 2001 έως το 2007 ανά τον κόσμο είχαμε 1440 ατυχήματα περίπου ε, και 356 πετρελοκυλίδες. Είχαμε ένα μεγάλο ατύχημα και σε αμερικανικά υδατά το 88 στη Νέα Σκοτία ε, με το θάνατο 167 ατόμων. Ο κύριος Ζήπερ είπε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη νομοθετική ρύθμιση η Αμερική σε σχέση με μας. Μα από το 2001 και μετά ισχύει απαγόρευση για τις υπεράκτιες εξορίξεις πετρελαίου ε, για το 85% της παράκτης περιοχής, ε, των παράκτιων περιοχών τον είπα. Μπορούμε να το συζητήσουμε με την Επιτροπή και τους συναδέλφους. Η Επιτροπή, ας πούμε, σκέφτεται μια τέτοια απαγόρευση για την υπεράκτια εξόρυξη πετρελαίου. Το να πούμε ότι δεν μπορούμε να λάβουμε μέτρα μέχρι να γνωρίζουμε τα επαρκή αίτια του ατυχήματος, ενώ τόσες, τόσες χιλιάδες ατυχήματα ε, έχουν συμβεί τα τελευταία 7 χρόνια. Πολλά ατυχήματα σημειώνονται κάθε χρόνο προφανώς υπάρχει πρόβλημα ε, με την ε, υπεράκτια εξόρυξη και πρέπει να ε, ληφθούν μέτρα. Πρέπει να αρχίσουμε τη συζήτηση γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι και μια τέτοια απαγόρευση έχει ενδεχομένως σοβαρότατες συνέπειες. Ευχαριστούμε η κυρία Κορίν Λεπάς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ τον ε, ε, Διευθυντή της ε, ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ Ενέργειας για τις εξηγήσεις που έδωσε. Η ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Πολιτικής πρέπει να ε, συμμετάσχουν στη συζήτηση, γιατί δεν τίθεται μόνο θέμα ε, εξέδρας, εξόριξης, ε, μιλάμε για σοβαρές επιπτώσεις και στο περιβάλλον και σε διάφορες άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Σε τρία επίπεδα νομίζω πρέπει να τοποθετήσουμε τον προβληματισμό μας. Πρώτον, ε, για την νομοθεσία ως προς την αδειοδότηση της εγκρίσης. Δυστυχώς ε, δεν ε, θα συμφωνήσω με τον ενθουσιασμό σας ότι υπάρχουν πολλά εφαρμοστά ευρωπαϊκά νομοθετήματα στον τομέα αυτό. Δυστυχώς δεν ισχύει αυτό. τα κείμενα που σχετίζονται με το πακέτο Έρικα δεν ισχύουν γιατί δεν μιλάμε για σκάφη, για πλοία. Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη δεν είμαι σίγουρη ότι είναι εφαρμοστέα σε αυτό το τομέα, οπότε αρχίζουμε να διαβλέπουμε ποια είναι τα αίτια ε, χοντρικά, όχι, χωρίς να ε, τα καταλογίσουμε όλα στην BP, ε, αλλά διαβλέπουμε τα αίτια και νομίζω ότι καλύτερα είναι να λειτουργήσουμε προώρα παρά με καθυστέρηση. Δηλαδή να δούμε τι μπορεί να συμβεί, όχι μόνο τι συνέβη. Ας αντλήσουμε τα διδάγματα μας από το παρελθόν, ναι μένα, αλλά ας δούμε και τι θα συμβεί στο μέλλον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ισχύους εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία για αυτό το τομέα, κυρίως για την αδειοδότηση. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να προβληματιστούμε, γιατί υπάρχει η εθνική νομοθεσία, ε, το νορβηγικό και το αγγλικό δίκαιο συγκεκριμένα. Έτσι, αυτά διέπουν την αδειοδότηση. Τώρα, δεύτερον, ε, το θέμα τη ευθύνη. προφανώς είναι ε, πολύ σημαντικό το ζήτημα και τη χάνει διαφορετικής μεταχείρισης ε, στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη αντίστοιχα. Ε, και αυτό οδηγεί σε διαφορετικέ συμπεριφορέ στον οικονομικό τομέα. Αν διατρέχετε σοβαρό κίνδυνο, σα αποδοθεί ευθύνη και γι' αυτό μιλάμε έτσι για τη ρήπανση, παραδείγματο χάρη με τα καύσιμα από τα πλοία. Αν λοιπόν διατρέχετε σοβαρό οικονομικό κίνδυνο, τότε λαμβάνετε όλα τα πετούμενα μέτρα ασφαλεία. Αν οι οικονομικοί φορεί όμω δεν διατρέχουν τέτοιο σοβαρό οικονομικό κίνδυνο, δεν αναλαμβάνουν αυτά τα μέτρα ασφαλεία. Είναι τόσο απλό. Ω εκ τούτου, ναι, να το σκεφτούμε αυτό που είπατε, αλλά δεν μπορεί να μην αποδοθεί καμία ευθύνη στους οικονομικούς φορείς για ε, τα ε, λάθη που διέπραξαν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας ε, της εξέδρας. Δηλαδή η BP συνέχισε να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο την εξέδραση στον κόλπο του Μεξικού και νομίζω ότι είναι αντιπαραγωγικό να μην αποδώσουμε καμία ευθύνη στην BP. Αφήστε που υπάρχει και το θέμα της εποπτείας. Ωραία να έχουμε τα νομοθετήματα Είπατε ότι είναι αυστηρή η Αμερικανική νομοθεσία. Εγώ δεν είμαι πεπισμένη πάντως. Ο πρόεδρος Ομπάμα τρεις εβδομάδε. πριν το ατύχημα είχε σκεφτεί να ε, υιοθετήσει αυστηρότερη ε, νομοθεσία και ανέβηκαν όλες τις επάλκε. Όχι, όχι, τα ελέγχουμε όλα, ε, δεν χρειάζεται περαιτέρω ρύθμιση. Μα δείτε στην πράξη τι συμβαίνει. Αυτό είναι που έχει σημασία και αυτό, αυτή η σκέψη μας οδηγεί σε μια άλλη σφαιρικότερη σκέψη που μας απασχολεί συχνά στην Επιτροπή μας, δηλαδή σταδιακά πώς θα κάνουμε για να ε, διαφύγουμε από αυτήν την κοινωνία του πετρελαίου, γιατί περί αυτού πρόκειται αφήστε που υπάρχει ένα επιπρόσθετο στοιχείο. Δηλαδή, στο μέτρο που ε, μειώνονται τα κοιτάσματα και τα αποθέματα, ε, και, ε, κατευθυνόμαστε το λένε και περισσότερο προς τις υπεράκτιες εξέδρες, μετά θα έχουμε την ασφαλτούχο, άμμο και άλλα τέτοια καύσιμα, τα αέρια του θερμοκηπίου κτλ. Οπότε αυτό είναι το θέμα που τίθεται. Μία μεταβατική λύση για να ξεφύγουμε από αυτή την κοινωνία κατανάλωσης πετρελαίου, γιατί αυτό που συμβαίνει στον κόλπο του Μεξικού. Ε, σε αυτή τη σκέψη πρέπει να μας οδηγήσει, δηλαδή οι οικονομικές και συνέπειες για την εταιρεία BP είναι σημαντικές. Οι αξιολογήσεις του κόστους ε, κυμαίνονται σήμερα από 19-49 δις δολάρια, ένα αστρονομικό το ποσό. Ε, θα πώς ε, θα ανταπεξέλθει η εταιρεία BP, θα μπορέσει. Ε, βλέπουμε ότι ήδη δεν μπορεί να συγκεντρώσει 20 δις για το Ταμείο Αλληλεγγύης. Αφήστε που εξετάζετε το ενδεχόμενο των 50 δις. Και δεύτερον, ε, πώς θα επηρεαστεί γενικότερα η οικονομία του πετρέλαιου. Και πανέρχομαι στο θέμα τη Ευθύνη, που σχολίαζα προηγουμένως, γιατί προφανώ μπορεί η βιομηχανία ε, πετρελαίου να θέλει να συστήσει αυτό το ταμείο, όπως ε, το ταμείο που υπάρχει για τις ε, καταστροφές που προκαλούν τα πλοία, για να πούνε ορίστε, απεκδιόμεθα τις ευθύνες, δεν θα αναλάβουμε εμείς την οικονομική ευθύνη που προκύπτει από την εξόριξη πετρελαίου, στο μέτρο που θα υπάρχει αυτό το ταμείο το οποίο θα μπορούσε να εγγυηθεί, να δώσει κάποιες εγγυήσεις για τα θύματα και να καλύψει το κόστος. Λοιπόν, ε, ε προεδρεύω με παράκτη περιοχή και αύριο θα εκπροσωπηθούμε σε μια ακρόαση που θα γίνει αύριο το ε, μέχρι τις 12.30. Θα υπάρξει και εκπρόσωπος της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ενέργειας, εκπρόσωποι από τον κλάδο και από μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Θα συζητηθεί το ε, θέμα της κείμενης νομοθεσίας και τα μέσα για τον έλεγχο και την την πρόληψη της ρήπανσης που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Στάς και ο Μισελ Ριμπασί μετά. Eh, eh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να πω ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε η συνάδελφος Λεπάζ συνόψισε με πάρα πολύ καλό τρόπο τις βασικές μου ανησυχίες. Θεωρώ ότι οι κρίσεις μπορεί να έχουν και θετικά αποτελέσματα. και εμείς εδώ αντιμετωπίζουμε κρίση. Η καταστροφή ε, στον κόλπο του Μεξικού θα μας επιτρέψει να εξαγάγουμε διάφορα συμπεράσματα. Καταρχάς, ε, οι πετρελαϊκές επιχειρήσεις δεν θεωρούν ότι είναι ε, ικανή και αναγκαία συνθήκη η ασφάλεια. Έχουν επιλέξει να κάνουν ακραίες εξορίξεις και στην πράξη δεν έλαβαν υπόψη τους πολύ σοβαρά τα θέματα της ασφάλειας. Τα τελευταία χρόνια, για να μπορέσουμε να κάνουμε και μία σύγκριση των στοιχείων, δαπανήθηκαν περίπου 39 δις δολάρια για την ε, ανακάλυψη νέων πηγών, νέων κοιτασμάτων και περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια για την έρευνα σε θέματα ασφάλειας. Τα στοιχεία νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχει την πρόθεση να εξαγάγει κάποια διδάγματα από τα όσα συνέβησαν στην Αμερική. Μήπως σκοπεύετε να ζητήσετε μια ανεξάρτητη έρευνα για θέματα ασφάλειας σε πετρελαϊκές πλατφόρμες ε, στα ευρωπαϊκά είδατα. Καλό θα ήταν να έχουμε μια ανεξάρτητη μελέτη για να γνωρίζουμε λίγο καλύτερα πώς έχουν τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εισαγωγή της μας είπε ότι ναι, υπάρχει πάρα πολύ ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Λεπάς. Ναι, έχουμε πάρα πολύ νομοθεσία, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα της νομοθεσίας προέκυψε μετά από την καταστροφή στο Έρικα και στο Πρεστής και βασικά αναφέρεται στην ρήπανση η οποία προκύπτει από τα πετρολοφόρα σκάφη και όχι από τη μόλυνση που έχουμε από πετρελαϊκές πλατφόρμες. Στις 7 Ιουλίου θα γίνει μια συζήτηση στην Ολομέλεια επί του θέματος. Μήπως ε, θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τη δέσμευση να παρουσιάσει στην αίθουσα της Ολομέλειας ε, το σύνολο της νομοθεσίας που ισχύει για τις πετρελαϊκές ε, εξορίξεις, γεωτρήσεις και τις πλατφόρμες προβλέπεται συζήτηση για τις 7 Ιουλίου και έτσι οι προβουλευτές θα μπορέσουν να έχουν μια ενημέρωση για το τι ισχύει και τι δεν ισχύει σε θέματα πετρολαϊκών πλατφόρμας. Ε, μετά, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια της Θάλασσας. Πρόκειται για έναν οργανισμό πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, έχει προκύψει από την ε, Λισαβόνα και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Όποιος όμως διαβάσει τον κανονισμό της ΕΜΣΑ γνωρίζει ότι η ΕΜΣΑ δημιουργήθηκε μετά από τις καταστροφές οι οποίες προκάλεσαν την ε, μόλυνση των υδάτων. Εκεί είχαμε ευθύνη από τα πετρολεοφόρα. Δεν έχει όμως συμπεριληφθεί το θέμα της, ε, του ενδεχομένου ε, μόλυνσης από πλατφόρμες. Ίσως θα μπορούσαμε λοιπόν να επεκτείνουμε την εντολή της ΕΜΣΑ, ώστε η τεχνογνωσία που διαθέτει δικαίως η ΕΜΣΑ να επεκταθεί και στα θέματα τα οποία προκύπτουν από καταστροφές, από τέτοια φαινόμενα, πετρελαϊκές πλατφόρμες. Ένα άλλο ερώτημα τώρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε προβλέψει κάποια στρατηγική, γνωρίζετε τι πρέπει να γίνει αν αντιμετωπιστεί μια πραγματική κρίση ρήπανσης από πετρέλαιο. Υπάρχει μια στρατηγική για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχουν κάποια σχέδια εκτάκτου ανάγκης από πλευρά ΕΜΣΑ. Οι συνάδελφοι Αρσένης και Λεπάζ είπαν ότι υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες ευρωπαϊκά ύδατα. Και το μεγαλύτερο τμήμα της διαχείρισης το έχει η Νορβηγία. Τι γίνεται σε θέματα συνεργασίας με την Νορβηγία. Μήπως θα έπρεπε να γίνουν κάποιες επαφές με τις νορβηγικές αρχές ώστε τα μέτρα τα οποία προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι συντονισμένα με την Νορβηγία. Κατόπιν, βοήθεια σε όσους πλήττονται από την ε, μόλυνση. Πρέπει να πω ότι διαπίστωσα με έκπληξή μου ότι σε απάντηση των καταστροφών του Έρικα και του Πρεστής, είχε προβλεφθεί να δημιουργηθεί ένα ταμείο για την αποζημίωση από την πετρελαϊκή ρήπανση στη θάλασσα και υπήρχε και μία πρόταση της Επιτροπής ε, το Δεκέμβριο του 2000 είχε συζητηθεί σε πρώτη ανάγνωση τον Ιούνιο του 2001 κατόπιν ε, τον Ιούλιο του 2002 ε, παρουσιάστηκε μια πρόταση αναθεώρησης και από τότε τα πράγματα έχουν μείνει στάσιμα. Γιατί δεν δημιουργήθηκε τελικά αυτό το ταμείο. Και εάν σε μια επόμενη θητεία ε, και ανάγνωση επεκταθεί η, η εντολή αυτού του ταμείου, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε αποζημιώσεις και για τέτοιου τύπου καταστροφές. Άνω του 15% των ε, εξεδρών ε, γεώτρησης ε, είναι άνω των 20 ετών. Κάποιοι από αυτούς είναι σε φάση παροπλισμού, κάποιες δηλαδή εξέδρες είναι πάρα πολύ παλιές και πρέπει να παροπλιστούν και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα πλατφόρμας. Αν κάτι δεν πάει καλά, ο κίνδυνος ε, μόλυνσης είναι τεράστιος. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω και για το σημείο αυτό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει κατά πόσον έχει εξετάσει το ενδεχόμενο ή σκοπεύει να εξετάσει το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποιες στρατηγικές για το μελλοντικό παροπλισμό αυτών των πετρελογικών εξεδρών και πώς μπορούμε να υποχρεώσουμε τις επιχειρήσεις ε, να αναλάβουν τις ευθύνες τους από οικονομικής πλευράς, διότι πραγματικά θεωρώ ότι είναι δική τους ευθύνη το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. και Σιμανή και κατόπιν κ. Παζέκατ. Ευχαριστώ την Επιτροπή που οργάνωσε αυτή την ε, ακρόαση. Γιατί έχω να πω ότι έχουμε τεράστιες ε, προβλήματα να πάρουμε τις από τον ίδιο τον επιτρολικό κλάδο. Ο βοηθό μου τηλεφώνησε παντού και όλο του είπανε θα σας απαντήσουμε αργότερα. Η δική μου ερώτηση είναι πολύ απλή. Υπάρχουν 27 πλατφόρμες ε, πεταλικής εξόρυξης στην Βόρειο Θάλασσα. Πρώτη ερώτηση. Ένα δυστύχημα σαν αυτό που έγινε στο ε, κόλπο του ε, Μεξικού θα μπορούσε να λάβει χώρα και Εάν έχουμε το ίδιο δυστύχημα, τι έχουν προβλέψει οι πετρελαϊκές εταιρείε. Γιατί τώρα μου λένε ότι δεν είχε προβλέψει, προβλεφθεί κάτι τέτοιο στα 1500 μέτρα. Δεν είχε προβλεφθεί ότι με αυτή την ε, ε, πίεση θα μπορούσαν να υπάρχουν οπωσδήποτε προβλήματα. Και έχουμε τώρα ακροές ε, δύο μήνες μετά. Εμένα μου λένε τώρα δεν είναι τόσο σοβαρό γιατί έχουμε ένα μέσο όρο 100 χρονομέτρων. Το 1999 στο κόρφο μουσικό είχαμε μία έκρηξη της πλατφόρμας Xtox 1 και χρειαστήκανε 10 μήνες για να κλείσει. Σε 50 μέτρα ήταν τότε αυτό. Δεύτερο της στιγμήματα. το 2009, στο Τιμόρ, στη θάλασσα του Τιμόρ. Η πλατφόρμα εξόρυξης ε, ήταν θύμα μιας εκρηξής πετρελαίου. Πού 80 μέτρα βάθος. Και χρειάστηκαν τρεις μήνες για να κλείσει. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι 25 πλατφόρμες που έχουμε, εκτός από ότι παλιώνουν, δεν έχουμε καμία εγγύηση ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Εσείς ρωτήσατε τους εκπροσώπους του κλάδου να πείτε έχετε τη δυνατότητα για να κλείσετε αν υπάρχει κάποιο ρήγμα και να υπάρχει έτσι μια εγγύηση ή δεν έχετε, θα πρέπει να σταματήσουμε το σύστημα λοιπόν. Δεύτερο, κάτι που με ανησυχεί. Ποιο τις ελέγχει τις πλατφόρμες αυτές. Ελέγχθη ότι η υπηρεσία που συνήθως ελέγχει τα σκάφη και τις πλατφόρμες, τις κινητέ πλατφόρμες, δεν ελέγχει τις πλατφόρμες offshore. Θα πρέπει λοιπόν να ζητηθεί διεύρυνση των ε, αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας αυτής ε, για να ελέγχουν οι λεκτές. Γιατί ποιος δίνει τις άδειες, τα κρατημέλη. Αλλά ίσως υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της, εκείνων που δίνουν τις άδειες και των εκπροσώπων του κλάδου. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει δηλαδή από την έμψα ο ελεγκτής των εθνικών ελεκτών. Και τελευταίο που με ανησύχησε είναι το αίτημα της Ιρλανδίας που ζήτησε να εγκαταστήσει μια πλατφόρμα σε 3.000 μέτρα βάθος. Βλέποντας τι γίνεται, ρωτάω στους συναδέλφους, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα μορατόριο. Δηλαδή να ζητήσουμε καταρχήν τις ε, Πρώτο δώσουμε στην Ολλανδία την άδεια για να κάνει μια εξόρυξη 3.000 μέτρα. Όσο ξέρουμε ότι στη 1.500 δεν μπορούμε να σταματήσουμε ε, σε περίπτωση που υπάρχει μια έκρηξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε για την περίληψη που μα έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλε τι ισχύουσε οδηγίε και τι δράσει που έχει αναλάβει αλλά δυστυχώς ε, δεν ικανοποιήθηκα με την παρατήρηση ότι ξέρουν ήδη τώρα πως ισχύουν πολλές οδηγίες, είναι εφαρμοστές πολλές οδηγίες, μα ε, δεν ισχύει αυτό. Ας πάρουμε ένα ζήτημα που θα μου πείτε ότι είναι απλό. Απόδοση ευθυνών στις πετρελαϊκές εταιρείες όταν κάτι πάει στραβά. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη. Το 1999 με την καταστροφή του ΕΡΙΚΑ τι μάθαμε ότι έπρεπε να προσαρμόσουμε την νομοθεσία μας, ε, πακέ, τα πακέτα ΕΡΙΚΑ έτσι για να ε, αποδοθεί ευθύνη για την μεταφορά πετρελαίου με πετρελαιοφόρα έπρεπε να κάνουμε αυτή την προσαρμογή. Οπότε τα πετρελαιοφόρα τώρα ε, έχουν ευθύνη, αλλά όχι οι εξέδρε εξόρυξη πετρελαίου. Λέει η Επιτροπή ότι πρέπει να διερευνήσει όλε τι οδηγίε, πρέπει να διερευνήσει τα αίτια του ατυχήματο στον κόλπο του Μεξικού. Ωραία. Για την ευθύνη δεν χρειάζεται να ξέρω τα αίτια. Ξέρω να ξέρω, αν ισχύει, θέλω να ξέρω αν ισχύει η αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Ε, ε, η μόνη οδηγία που επηρεάζει τον κλάδο είναι η οδηγία περί Σα ευθύνης. Σας παραπέμπω σε αυτή την οδηγία. σαφώ αναφέρει ότι οι εταιρείε φέρουν ευθύνη μόνο αν ε, υπάρχει αντίκτυπο στα ύδατα βάσει τη οδηγία πλαισίου για τα ύδατα ή στο έδαφο ή στη βιοπικιλότητα βάσει της οδηγίας ε, για, τα, για τους βιοτόπους. Ωραία. Τώρα ξέρουμε ότι έχουμε και οδηγία ε, για τα ορυχεία και εκεί βλέπουμε τις απαιτήσει ε, απειλή προς την ανθρώπινη ζωή για το περιβάλλον ε, με την ευρύτερη έννοια. Αυτό όμως δεν ισχύει στην οδηγία περιβαλλοντικής ευθύνης αν κάτι πάει στραβά στις εξέδρες εξόριξης πετρελαίου. Μία απλή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν ε, προετοιμάζεται επέκταση της ε, τωρινής οδηγίας ε, περιβαλλοντικής ευθύνης και να καλύπτει τις γενικές απειλές για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον και την προστασία των υδατών ή στην αναθεώρηση θα ασχοληθείτε μόνο με τις πετρελαϊκές εξέδρες. Θα ήθελα μια απλή απάντηση σε αυτή την απλή ερώτηση που κάνω. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ κάποιες παρατηρήσεις και μετά θα πάρει το λόγο ο Πίτερ Λίζε. Το Μάιο υπέβαλα ένα σχέδιο ψηφίσματος που απερίφθη δυστυχώς από τη διάσκεψη των Προέδρων. Παρόλα αυτά όμως οδήγησε σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Στρασβούργο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα το ταχύτερο δυνατόν και να εγκρίνουμε ένα ψήφισμα για αυτό το θέμα. Ο συνομιλητής μας είναι ένας εκπρόσωπος από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ενέργειας, όπως και στο Στρασβούργο αλλά εμείς θα θέλαμε να αναλάβει σημαντικότερο ρόλο επίτροπος αρμόδιος για τα θέματα περιβάλλοντος. Δεν είναι θέμα βιομηχανίας, δεν είναι μόνο ενεργειακό το ζήτημα. Σαφώς ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια περιβαλλοντική διάσταση. Η γάμα δέλτα ενέργειας θα πρέπει να υποχωρήσει για να αφήσει την Επίτροπο αρμόδια για τα περιβαλλοντικά θέματα να ε, έλθει στη σκηνή. Η Επιτροπή αγνόησε την έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις περιβαλλοντικές ε, συνέπειες ε, της οικοδόμησης του Αγούρ Nord εμείς εγκρίναμε την έκθεση και δεν έκανε απολύτως τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για ποιο λόγο αναρωτιέμαι. Σε πολλές περιπτώσεις νομίζω ο λόγος είναι ότι είναι ισχυρότερο το βιομηχανικό λόμπι σε σχέση με το περιβαλλοντικό ε, λόμπι, με τις περιβαλλοντικές ομάδες ε, πίεσης. και αποσιωπούμε τα περιβαλλοντικά θέματα επειδή υπάρχει αυτό το ισχυρό βιομηχανικό λόμπι. Λοιπόν, απευθύνω έκκληση ε, στην ε, ε, ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Περιβάλλοντος να αναλάβει σημαντικότερο ρόλο. Σημειώθηκαν πάρα πολλά ατυχήματα στη Βόρεια Θάλασσα 32 ατυχήματα όπου χρειάστηκε να σφραγιστεί η υποθαλάσσια πετρελαιοπηγή από τις 103 ε, υπεράκτης ε, εξέδρες που υπάρχουν. και που διανύχθηκαν το 70, ε, οι 47 έχουν ακόμη προσδόκιμο ζωής 5 ε, ετών και οι 23 έχουν ήδη υπερβεί το, την ωφέλιμη ζωή τους ε, και τεχνητός πώς έχει παραταθεί η διάρκεια ζωής τους. Σε αυτά τα 30 τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικότατες τεχνολογικές εξελίξεις και χρειάζεται αναθεώρηση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την ιδέα εξαγοράς ε, του χρόνου μέχρι να δούμε ε, τι οδήγησε σε αυτή τη συγκεκριμένη έκρηξη. Είναι πάρα πολύ απλό έχετε την ε, θάλασσα, έχετε τα ειζήματα πετρελαίου μέσα στη θάλασσα και έχετε τον αγωγό που συνδέει τα κοιτάσματα με την επιφάνεια. Ωραία. Χρειάζεστε έναν αγωγό που δίνει τα μέγιστα ηχέγγυα ασφαλείας και χρειάζεται και ένας ε, μηχανισμός παρακολούθησης, εποπτείας. Αν τώρα προσπαθείτε να εξοικονομήσετε χρήματα, ναι, θα, τελικά θα πληρώσετε 20 δις για αποζημίωση. Όμως, τι γίνεται όταν συμβαίνει αυτό σε ένα φτωχότερο μέρο του κόσμου, στην Αφρική, όπου κανείς δεν αποζημιώνεται για τέτοια ατυχήματα. Πίτερ Λίζε, παρακαλώ. Και Λίντα Μακέβαν, κάτω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Κουκουσλάφ, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπες μόλις τώρα Καταρχήν, ευχαριστώ τον Ρίχαρτ Τζέιμπερ που έθεσε το θέμα αυτό στην μεσαία διάταξη γιατί απασχολεί όλους τους πολίτες στην Ευρώπη και θα πρέπει να εξετάσουμε και τις συνέπειες. Η πιο σημαντική συνέπεια για μένα είναι αυτό που είπε και η Κορίν Λετάζ και που είπε και την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος Ομπάμα. Υπάρχει συμπληρωματικό επιχείρημα να μειώσουμε την εξάρτηση από το πετρέλαιο και να χρησιμοποιήσουμε περισσότερε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Και ελπίζω αυτό το έχουμε πάντα κατά νου όταν συζητάμε τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Αυτό που είναι σημαντικό βέβαια είναι ότι στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε πιο αυστηρές διατάξεις για το ένα από ότι για το άλλο γιατί όταν συζητάμε για τα βιοκαύσιμα δημιουργώ την εντύπωση ότι ζούμε σε ένα ειδικό κόσμο και μέχρι στιγμής δεν χρειαζόμαστε καθόλου ενέργεια και τώρα ξαφνικά έχουμε τα βιοκαύσιμα. Όχι. Κάθε ένα λίτρο βιοκαυσίμων που παράγεται αντικαταστά ένα λίτρο πετρελαίου. Και εάν ένα πετρελαιοφόρο με βιοκαύσιμα να βαγίσει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει για το κάδμιο στη φωτοβολταϊκή, για την αιωλική ενέργεια και τα πτηνά. Όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι κίνδυνοι πολύ πολύ μικρότεροι από εκείνοι που προέρχονται ή που μπορούν να προέλθουν από το πετρέλαιο. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου. Κάποιε συγκεκριμένε ερωτήσει τώρα προ την Κομισιόν. Ο πρόσωπο τη Κομισιόν είπε ότι στα ευρωπαϊκά ύδατα το βάθος εξόρυξης είναι μικρότερο. Δεν κατάλαβα όμως ακριβώς. Καταρχήν ελέγχθη κατά μέσο όρο 90 μέτρα και μετά κατάλαβα ότι πάει μέχρι 200 μέτρα, μετά ότι πάει μέχρι 700 μέτρα. 700 μέτρα βέβαια είναι σημαντικό βάθος όπου οπωσδήποτε δεν είναι πολύ εύκολο να ε, βουλώσει κανείς κάποιες, ε, κάποια προβλήματα που υπάρχουν. Και υπάρχει επίσης και μία πληροφορία που αφορά τις εξορίξεις της ΜΠΕ στα νησιά Σέτλαν στα 400 μέτρα. Αυτό τι σημαίνει, η κατάσταση παρόμοια με εκείνη του κόλπου του Μεξικού ή μπορούμε να αποφύγουμε καταστροφές. Δεύτερον, θα ήθελα να ξέρω ακριβώς τον αριθμό των πλατφόρμων εξορίξης στη, στα ευρωπαϊκά ύδατα. Η κυρία Ριβαζή αναφέρθηκε σε 27. Εγώ από τις γερμανικές υπηρεσίες άκουσα 450 πλατφόρμες στη Βόρεια Θάλασσα. Υποθέτω ότι οι υπηρεσίες της Κομισιόν έχουν το ακριβό στοιχείο που θα μπορούσαν να μας δώσουν. Η νορβηγική κυβέρνηση εισήγαγε μορατόριο για βαθιές εξορίξεις. Τι θα πει βαθιές. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει κανένας. Αυτό θα ήθελα να μου το πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μετά να αναφερθώ σε αυτό που ανέφερε ο Μπασέκο. Το θέμα της ευθύνης για περιβαλλοντικά προβλήματα. Παρακολούθησα πολύ προσεκτικά το θέμα, όταν συζητάγαμε το θέμα τη ευθύνη όπου δεν ήταν επί τη ουσία αρμόδια η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αν θυμάμαι καλά, για τα διεθνή ύδατα... Και τι πλατφόρμε αυτέ τα διεθνή ύδατα, συγγνώμη, τι είχαμε αποκλείσει, γιατί είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν γι' αυτό διεθνεί συμβάσει. Αλλά ξέρουμε, αν περιμένουμε για διεθνεί συμβάσει, θα περιμένουμε πολλέ φορέ 20 χρόνια. Λοιπόν, η συγκεκριμένη μου ερώτηση είναι η διεθνή κοινότητα πόσο έχει προχωρήσει στο διαγωνισμό. Εγώ δεν έχω υπόψη μου καμία διεθνή σύμβαση για την περιβαλλοντική ευθύνη στην ανοιχτή τα θάλασσα, ούτε για τις πλατφόρμες εξόρυξης, ούτε για τα πετρελαιοφόρα. Δεν θα μπορούσε γλίγορα να προχωρήσει η Κομισιόν να υπάρχει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακέβεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και σένα Μπογκοσλάβ διότι εσύ ήσουν αυτός που έθεσε το θέμα αυτό πριν από κάποιες εβδομάδες και είπε ότι πρέπει να πάει στην Ολομέλεια και εγώ τότε είχα πει ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. δεν με ενοχλεί τόσο πολύ να βρίσκεται στην Ολομέλεια, αλλά το να έχουμε ψηφίσματα βεβιασμένα ορισμένε φορέ δεν είναι σωστό. Ορισμένε φορέ πιαζόμαστε στο κοινοβούλιο γιατί θέλουν όλοι να έχουν δελτία στον τύπο, ενώ καλό θα ήταν να περιμένουμε και να το συζητήσουμε ορίστε. Το συζητάμε στην Επιτροπή τώρα. Άκουσα τόσα διαφορετικά στοιχεία για το πόσες πλατφόρμες έχουμε στην ε, Βόρεια Θάλασσα, πόσο παλιές είναι. Δεν ε, είναι σαφές και το βάθος, ε, ποιο είναι το βάθος, το μέγιστο επιτρεπόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γίνεται, εθνικό δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο, ποιο αποφασίζει. Ε, νομίζω αποφασίζουμε σε εθνικό επίπεδο, αλλά υπάρχει καθοδήγηση από ε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, καλό θα ήταν λοιπόν να μας δώσετε κάποια στοιχεία, να ξέρουμε πόσες πλατφόρμες έχουμε, τι ηλικία έχουν, ε, τι βάθος έχουν, πόσο μακριά απέχουν από τις ακτές, όλα αυτά τα βασικά θέματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε και να κατανοούμε. Είμαι βέβαιη ότι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, αλλά είναι δύσκολο να τις βρω όλες μαζεμένες. Και χρειαζόμαστε και κάποια στοιχεία για το ποιο είναι υπεύθυνο γιατί. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, εξ όσων κατάλαβα, υπάρχουν ε, διαδικασίε λήψη αποφάσεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο για τι εξορέξει πετρελαίου και όλα σχετίζονται από την απόσταση από την ακτή. Ε, εξετάζουν μια προηγούμενη ενημέρωση πριν από την πετρελοκυλίδα Κάποιο υπεύθυνο στι ε, Τρία μίλια θεωρείται απόφαση ομόσπονδου ε, κράτους, ενώ πάνω των τριών μιλίων είναι πλέον η ε, ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών. και θέλουν να δώσουν στις πολιτείες μεγαλύτερο έλεγχο στις ε, εξορίξεις ε, και αυτό νομίζω ότι είναι και η κατεύθυνση που θέλουν να ακολουθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, κάποιος είπε και για τη συζήτηση που θα κάνουμε στην Ολομέλεια, κάποιος είπε ότι θα γίνει 9 η ώρα το βράδυ στις 7 Ιουλίου. Είναι σημαντική αυτή η συζήτηση και 9 η ώρα το βράδυ της Τετάρτης ε, δεν είναι η καταλληλότερη ώρα. Ε, πριν όμως γίνει συζήτηση, είμαι βέβαιη ότι θα έχετε κάποια στοιχεία να μας δώσετε. Είμαι βέβαιη ότι έχετε ετοιμάσει κάποια στοιχεία για τους επιτρόπους και θα θέλαμε να μας τα δώσετε και εμά για να είμαστε ενημερωμένοι και εμείς. Θα ήθελα να μου πείτε επίση, να μου απαντήσετε βασικά τι ερωτήσει που ακούσαμε. Ακούσαμε διάφορα στατιστικά στοιχεία για το βάθο. Είναι τα επιτρεπόμενα, είναι νομοθεσία, είναι η πάγια πρακτική. Υπάρχουν κάποια κράτη που δίνουν έγκριση για βαθύτερα ε, σημεία. Κάτι άκουσα τώρα για την Ιρλανδία, αυτή είναι η απόφαση του Ιρλανδικού κράτους. Σε τι κλίμακα βασίζεται, πώς γίνεται η απόφαση. Συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόλου σε αυτή την απόφαση. Και τέλος, νομίζω θα πρέπει να το συζητήσουμε και στη συνεδρία των συντονιστών δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς συνέβη στις ΗΠΑ και δεν θα πρέπει να καταλήξουμε σε βεβαιασμένα συμπεράσματα. Ε, αυτό που ξέρουμε είναι ότι όταν συμβεί κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το σταματήσουμε και τα αποτελέσματα είναι καταστρεπτικά. Επομένως θα πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα του ποιο πληρώνει. Το να είναι μια επιχείρηση που πληρώνει, ναι μεν καλό ακούγεται, αλλά αν χρεοκοπήσει η επιχείρηση τότε θα πληρώσει ο φορολογούμενος. Πρέπει να το δούμε λίγο μακρόπνοα, πρέπει να το συζητήσουμε και στην Ολομέλεια, αλλά χρειάζεται μια μακρόπνοη προοπτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας πείτε λίγο και πότε εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχετε συγκεντρώσει όλες σας τα αποτελέσματα ώστε να αποφασίσετε τι θα κάνετε. Υπάρχει μια καταληκτική προθεσμία τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο πριν από το τέλος του έτους που θα πείτε ότι ορίστε, τα έχουμε μαζέψει όλα και θα αποφασίσουμε τώρα τι κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Η Έλενα τον έσκου στη συνέχεια. και μετά ρατβίλε Μορκουνάιτε. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, και ευχαριστώ, κύριο Σέβερ, που μα έδωσε δυνατότητα να έχουμε την αλληλεγγύη αυτή απόψε με την ε, Κομισιόν. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπαν οι συνάδελφοι Σόνι και Ζίμπερ, που θέλουν να υπάρχει ψήφισμα του Κοινοβουλίου, γιατί το θέμα είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό η εκροή του πετρελαίου που ξεκίνησε τον Απρίλιο είναι μάλλον η μεγαλύτερη καταστροφή και όπως ο συνάδελφος Ζέμπα ήδη είπε θα μπορούσαν όλα αυτά να οδηγήσουν σε μια αλλαγή άποψη στις ΗΠΑ και στις άλλες χώρες. Και εμένα με ανησυχεί το θέμα του κινδύνου και θα πρέπει νομίζω η Κομισιόν να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για να μπορέσει να αξιολογήσει την κατάσταση ε, κατά πόσον γίνονται αυτές οι, ε, οι, οι έρευνες, αυτοί οι έλεγχοι στις πλατφόρμες και θα πρέπει να αξιολογήσουμε τους κινδύνους αυτούς σε ποιο βαθμό υφίστανται, γιατί ένας κίνδυνος 100% βέβαια δεν μπορεί να υπάρχει. Ε, μία η επιχείρηση πληρώνει το κόστος μιας τετοια πλατφόρμας που στην περίπτωση της BP ήταν ένα εκατομμύριο ε, την ημέρα και θα πρέπει γι' αυτό να εξασφαλίσουμε ο κίνδυνος των, των αυτών να μην ξεπερνάει το ενδεχόμενο κέρδος, γιατί στην περίπτωση αυτή βέβαια οι επιχειρήσεις δεν θα κάνουν ακριβώς ό,τι πρέπει. Έχουμε εδώ την τη μεγαλύτερη ε, επιχείρηση στον κόσμο, την BP, η, την οποία την ξεπερνάει το μέγεθος των ζημιών θα αναγκαστούν ε, πολλοί να πάρουν δάνεια για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ε, τις επιπτώσεις της καταστροφής. Όλοι θα θέλαμε να ξέρουμε βέβαια τι γίνεται εάν μια πιο μικρή επιχείρηση έχει την ευθύνη μια τέτοια περιβαλλοντολογική καταστροφή. Όπως ο κύριος Ζέμπερτ, έτσι και εγώ θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο δεν χρειάζεται να υπάρχει μία ομάδα ε, άμεσης κρούσης, μία task force για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών και θα ήταν καλό προσεχώς να μας υποβάλει νομοθετικές προτάσεις η Κομισιόν. Θα πρέπει να υπάρχουν και πιο αυστηροί όροι για την έγκριση αυτού του τύπου των ε, δραστηριοτήτων. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η κατάρτιση του προσωπικού. Γιατί βέβαια αυτές οι εξορρυκτικές ε, πλατφόρμες είναι διαφορετικές η μια από την άλλη και θα πρέπει η κατάρτιση του προσωπικού να είναι ανάλογη. Θα πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου τη, τους όρους των εκάστοτε συμβάσεων για να, μπορεί να, να μην μπορεί καμία επιχείρηση να κρυφτεί πίσω από τέτοιου είδους διατάξεις όταν υπάρχει κατά καταστροφή. Ευχαριστώ. Ρέντ Βίλε Μορκουνάιτε τώρα. και ο κύριο Παύλ Πότ στη συνέχεια και μετά εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστώ για την τόσο σημαντική αυτή συζήτηση τη καταστροφή ε, του κόλπου του Μεξικού. Αυτό άνοιξε σε πολλούς ε, τα μάτια Είχαμε ξαναζητήσει το θέμα των μηχανισμών ε, κάλυψης του, ε, των ζημιών. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν είναι σαφές ε, οι επιπτώσεις αυτού του τύπου της καταστροφής. Η ΜΠΠ κατηγορείται πλιστάκης, ε, αμφισβητούν τους συσχετισμούς όσον αφορά τις εγκρίσεις που έχουν δοθεί, την εκτίμηση των επιβεροντολικών επιπτώσεων. Πολλές φορές θεωρήθηκε μονομερής η αξιολόγηση αυτή. Ε, θα πρέπει λοιπόν ίσως να σκεφτούμε την αρχή της διαδικασίας και την εξολόγηση των επιπτώσεων για το περιβάλλον. Ίσως θα ήταν πιο απλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις μιας τέτοιας φυσικής καταστροφής. Βέβαια, οι μεμονωμένες επιχειρήσεις ε, έχουν πολύ πιο μεγάλα προβλήματα να αντιμετωπίσουν και οι Κομισιόν θεωρούν ότι τέτοιες ε, εταιρείε πετρελαιδών θα πρέπει να συνάπτουν μια ασφάλεια δεσμευτική. Γιατί όταν αναφερόμαστε σε χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτες χώρες, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μία πλατφόρμα εξόρυξης στην ε, Βαλτική θάλασσα που ε, ανήκει σε ρωσικές εταιρείε και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο υπάρχει κάποιος σχετικός διμερής διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσίας. Ευχαριστούμε, Ραντβίλε Παύλ Πότς. Η ερώτησή μου, πολύ σύντομα, έχει να κάνει με την ερυθρά θάλασσα. 160 χιλιόμετρα από τις Αιγυπτιακές ακτές είναι το Τζέρμπαν Αλσάιτ. Και εκεί, όπως και στον κόλπο του Μεξικού, αλλά σε μικρότερη κλίμακα, υπάρχει μια πετρελοκυλίδα. Δεν ε, αναφέρεται και πάρα πολύ στον τύπο, κυρίως γιατί είναι τουριστική περίοδος στην Αίγυπτο και επομένως η Αιγυπτιακή κυβέρνηση προσπαθεί να το αποσιωπήσει. Ε, τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιάννη Μπάνεκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη της Επιτροπής που εξέφρασαν τις απόψεις τους. οι ερωτήσεις είναι τόσες πολλές και τόσο διαφορετικές που ξέρω ότι όσο σκληρά και αν προσπαθήσω σίγουρα δεν θα μπορέσω να ικανοποιήσω τους πάντες. Θα προσπαθήσω όμως ε, να απαντήσω βάσει σημειώσεων που κράτησα. Αντί να απαντάω τη μία ερώτηση μετά την άλλη ή τον ένα ομιλητή μετά τον άλλο, ας ε, πάμε αναθεματική ενότητα. Καταρχάς ακούσαμε μία ερώτηση για το ποια νομοθεσία ισχύει, πού και ποιος αποφασίζει τι κλπ. οποιοδήποτε κράτος μέλος, ε, σύμφωνα με τις συνθήκες, με το πρωτεύον δίκαιο συμπεριλαμβανομένης και της συνθήκης της Λισαβόνας, δίνει στα κράτη-μέλη την απόλυτη κυριαρχία για τις ε, πηγές που θέλουν να εκμεταλλευτούν στην επικράτειά τους. Κάθε κράτος μέλος λοιπόν είναι αυτό το οποίο αποφασίζει πότε θα επιτρέψει οποιαδήποτε μορφή έρευνας, γεώτρησης ή παραγωγής ε, πετρελαϊκών πηγών στη χώρα τους αυτή τη στιγμή αποφασίσουν, υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που τους υποχρεώνει ε, η εκχώρηση αδειοδότησης και δικαιωμάτων να γίνεται κατά τρόπον ώστε να επιτρέπεται ισότιμη ε, συμπεριφορά ε, από όλους τους ευρωπαϊκούς φορείς που συμμετέχουν στο θέμα αυτό. Αυτή τη στιγμή δοθεί η άδεια ανεξάρτητα σε ποιον θα δοθεί, υπάρχει δέσμευση από την νομοθεσία για το κράτος μέλος να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσει καταρχάς για την απόκτηση της άδεια και κατά δεύτερον για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Η νομοθεσία αυτή είναι ε, συγκεκριμένος προς το εθνικό δίκαιο, δηλαδή υπάρχει εθνικός ε, ρυθμιστή ρυθμιστής σε κάθε κράτος μέλος, αλλά πολλά από τα όσα κάνει καθορίζονται από την εφαρμοστέ ευρωπαϊκή νομοθεσία γιατί ισχύουν αρκετοί νόμοι από αυτού. Ε, στη συζήτηση υπήρξαν πολλές επικρίσεις ότι δεν υπάρχει επαρκής νομοθεσία ε, και ζητήθηκαν και συγκεκριμένα παραδείγματα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα νομοθέτημα το οποίο καλύπτει όλες τις πτυχές ε, της διαδικασίας εξόρισης ε, γεώτρησης παραγωγής. Υπάρχουν κανόνες που διέπουν ε, την νομοθεσία που ισχύει για τις τεχνικές απαιτήσεις. Υπάρχει δηλαδή μια οδηγία η οποία καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις ε, για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, ε, το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε δυνητικά επικίνδυνο περιβάλλον, τι πρέπει να πληρείται σε αυτές τις περιπτώσεις, ε, τι πρέπει να πληρείται από θέματα ασφάλειας. Υπάρχουν λοιπόν οδηγίες οι οποίες πρέπει να μεταφέρονται σε εθνικό δίκαιο και πρέπει να πάμε και ακόμα περαιτέρω και να επιβάλλονται από εκεί και πέρα σε εθνικό επίπεδο. Πέραν αυτών, εκ παραλίλου, υπάρχει και άλλη νομοθεσία η οποία βασίζεται μεν τη Ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά υπό τη μορφή εθνικής ε, νομοθεσίας για τα θέματα της ασφάλειας και της υγείας ε, του προσωπικού που εργάζεται σε αυτέ τις πλατφόρμες. Επιπλέον υπάρχει και αρκετά εκτεταμένη νομοθεσία για ε, περιβαλλοντικές πτυχές αυτών των διαδικασιών. Ίσως θα έπρεπε να είχα πει ότι στην αρχή, όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει τι πηγέ θέλει να διαθέσει προς εκμετάλλευση, εάν βρίσκονται σε υπεράκτια υδατά, θα πρέπει οι αποφασίσεις να λαμβάνονται βάσει των υποχρεώσεων που καθορίζονται στην οδηγία για το ε, πλαίσιο της θαλάσσιας στρατηγικής. Πρόκειται για μια νέα νομοθεσία, η οποία, αν θυμάστε καλά, έγινε το 2008 και καθορίζει ένα ελάχιστο πλαίσιο εντό του οποίου τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές προκειμένου να έχουν μόνο ε, εποφελείς διαδικασίες στα υδατά τους. Πρόκειται λοιπόν για προϋπόθεση, έπρεπε να το είχα πει ε, εξ αρχής, ζητώ συγγνώμη που σας πάω προς πίσω, να πάμε τώρα μπροστά στην ίδια την επιχείρηση. Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα θέματα ασφαλείας ε, του προσωπικού καθώς επίσης και του περιβάλλοντος ε, διέπονται από συγκεκριμένα νομοθετήματα. Υπάρχει εθνική νομοθεσία αλλά σε μεγάλο βαθμό έχει προκύψει και διαμορφωθεί από οδηγίες που προέρχονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι την πρωτεύουσα ευθύνη για την ε, εποπτεία της συμμόρφωσης προς την νομοθεσία ε, την έχουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τα κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη έχουν μία εθνική ρυθμιστική αρχή, κάποιοι άλλοι τα έχουν ε, κατανεμημένα σε δύο-τρεις διαφορετικές υπηρεσίες, τα θέματα του περιβάλλοντος είναι αλλού, τα θέματα της υγείας είναι αλλού, άλλοι τα έχουν συγκεράσει σε ένα ρυθμιστή για τις υπεράκτιες δραστηριότητες η προσέγγιση διαφέρει. Ε, αλλά επειδή ακριβώς έχουμε κυρίως εθνική ευθύνη ρυθμιστών και αυτό φυσικά προκύπτει από το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα εκμετάλλευση των πηγών τους, θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη να συνεργαστούμε πιο εντατικά με τους εθνικούς ρυθμιστές και γι' αυτό ακριβώς τους καλέσαμε για την πρώτη συγκεκριμένη συνεδρίαση ε, για τις υπεράκτες δραστηριότητες που θα γίνει την Παρασκευή για να ξεκινήσει η διαδικασία συζητήσεων με τις εθνικές διοικήσεις προκειμένου να συζητήσουμε μαζί τους και να δούμε τι πρακτικές έχουν ε, χρησιμοποιήσει χωρίς να καταλήγουμε σε συμπεράσματα, αλλά έχουμε λάβει και κάποια μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε ότι ορισμένε φορές οι ρυθμιστές δεν έχουν τα πάντα έτοιμα, τουλάχιστον αυτά διαβάζουμε στον τύπο. Επομένως προκύπτει το εύλογο ερώτημα, διαφέρουν καθόλου οι εθνικοί ρυθμιστές, οι ευρωπαίοι ρυθμιστές. Γι' αυτό ακριβώς και τους έχουμε καλέσει όλους μαζί την Παρασκευή για να συζητήσουμε μαζί τους και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε ε, απόδοση στο μέγιστο δυνατό επίπεδο και για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και για την προστασία του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Όπως σας είπα, όση νομοθεσία και να έχουμε δεν θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε 100% ασφάλεια. Όλα αυτά προκύπτουν από μέγιστη συμμόρφωση, βέλτιστη επαλήθευση κτλ. Αλλά θα πρέπει πάντα να γνωρίζουμε ότι μπορεί να προκύψουν ε, δυστυχήματα και μπορεί να ε, προκύψουν δυσκολίες. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περιλαμβάνει κάποιες διατάξεις που καθορίζουν ποιος έχει την ευθύνη και καθορίζουν τα θέματα ευθύνης. Ακούσαμε πάρα πολλά για την οδηγία περιβαλλοντικής ευθύνης. Έχω μια νομική ανάλυση εδώ, σε μια μισή σελίδα, ε, περιγράφει πώς ισχύει η οδηγία περί παραβολαντικής Αυτό το ετοίμασαν οι συνάδελφοι στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Και εδώ μπορώ να σας πω ότι δεν ισχύει η δήλωση ότι δεν ισχύει η οδηγία περί παραβολαντικής ευθύνης. Επιπλέον όμως δεν θα είναι η μόνη οδηγία που θα ισχύει σε περίπτωση που έχουμε πετρελοκυλίδα από υπεράκτιες δραστηριότητε. Υπάρχει μια οδηγία γενική αποβλήτων η οποία εγκρίθηκε αρχικώς το 2006 αλλά αναθεωρήθηκε το 2008 και η αναθεώρηση τίθεται σε ισχύ το Δεκέμβριο του 2010 και αυτή η νομοθεσία θα καθορίζει σαφώς ότι ο ιδιοκτήτης του πετρελαίου, δηλαδή αυτός που έχει την άδεια, είναι ο υπεύθυνο για ζημίες που προκαλούνται όταν το πετρέλαιο δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Επιπλέον, όταν αξιολογούμε την κάθε νομοθεσία που ισχύει, είναι σημαντικό να μην δούμε μόνο την νομοθεσία αλλά και την ομολογία, δηλαδή από ποια υπόθεση έχει προκύψει κάτι. Ε, και εδώ έχουμε κάποιες δικαστικές ε, αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θέλουν να ενισχύσουν ε, περαιτέρω την εγκυρότητα της οδηγίας των αποβλήτων σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν δέχομαι λοιπόν τη δήλωση ότι η ευθύνη δεν καλύπτεται. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω την αρχική μου παρέμβηση που σας είπα ότι κάνουμε μια διεξοδική εξέταση της εφαρμοστέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εάν τυχόν καταλήξουμε στο συμπέρασμα, και αυτό δεν το κάνει μόνο η Γενική μου Διεύθυνση αλλά το, ε, ενεργείας, αλλά το κάνουν όλες οι Γενικές Διευθύνσεις που έχουν νομοθεσία ε, και κοινοτικό κεκτημένο που εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση. Εάν λοιπόν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει νομοθεσία που δεν καλύπτει επαρκώς ε, τα θέματα των υπεράκτιων δραστηριοτήτων, θα παρουσιάσουμε κατάλληλες πρωτοβουλίες. Μου ζητήσατε ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχει αυτή η μαγική ημερομηνία για την οποία θα σας δώσουμε τα στοιχεία. Καλό είναι να έχουμε συγκεκριμένους στόχους, πολύ ωραίο, αλλά θα πρέπει να τους θέτουμε και τους στόχους για να μπορεί κάποιος να τους χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς και από εκεί και πέρα να επιταχύνει αναλόγως, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε δράση μόλις προκύψουν αποτελέσματα. Η αναθεώρηση της κείμενης νομοθεσίας ε, γίνεται αρκετά γρήγορα η περιβαλλοντική νομοθεσία και η οδηγία περί περιβαλλοντικής ευθύνης είναι ήδη σε διαδικασία αναθεώρησης, κάτι το οποίο έχει έμεση επίπτωση στο σεβασμό του περιβάλλοντος, δεν έχει άμεση σχέση με, την, με τα όσα συνέβησαν στον κόλπο του Μεξικού, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει την εφαρμογή και να εξετάσει κατά πόσο μεταφέρθηκε σωστά η οδηγία και νομίζω ότι θα είναι έτοιμη σε κάποιους μήνες. Δεν ξέρω ακριβώς ποια ημερομηνία αυτή τη στιγμή. Και φυσικά θα ελέγξουμε και την οδηγία για θέματα ασφάλειας σε υπεράκτητε πλατφόρμες και επομένω θα έχουμε αποτελέσματα σύντομα. Μπορεί επίσης ε, να έχουμε και άλλε ε, αναθεωρήσεις νομοθεσίας, οι οποίες μπορεί να καθυστερήσουν λίγο περισσότερο κάποιε εβδομάδε ή και μήνε, αλλά όπως σας είπα, δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε με νέα νομοθεσία, αλλά αναφερόμουν σε οποιαδήποτε νέα νομοθεσία που θα καλύπτει κάποιες συγκεκριμένες ε, τεχνικές ε, απαιτήσεις, επί παραδείγματι. Ορισμένες φορές βλέπουμε ε, στον τύπο κάποιες ε, αναφορές ε, σε τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται ή δεν απαιτείται σε συγκεκριμένη νομοθεσία και νομίζω ότι δεν πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις επί τέτοιων θεμάτων εάν δεν διαπιστώσουμε ότι υπήρχε κάποιος ελληπής εξοπλισμός ή αν υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα το οποίο οδήγησε στο ατύχημα. Για την υπόλοιπη νομοθεσία όμως θα προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και θα παρουσιάσουμε πρωτοβουλίες. Ως προς τα αριθμητικά στοιχεία τώρα. Ναι, έχουμε στοιχεία για το πόσες ε, πλατφόρμες έχουμε. Έχουμε 123 πλατφόρμες στις οικονομικές ε, περιοχές ε, των ευρωπαϊκών χωρών. Εδώ έχουμε και την Ορβηγία δηλαδή. Και έχουμε και 148 πλατφόρμες γεωτρήσεων στην περιοχή. Δεν είναι όμως σωστή συζήτηση να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα νούμερο που θα δημιουργήσει και επιχαίους τίτλους. Δεν έχει σημασία ε, αν μιλάμε για κινητές ή για πλατφόρμες ε, Υπάρχει ένα σωρό εξοπλισμό που υπάρχει διαθέσιμο στα ύδατα. Δεν μιλάμε για ένα ενιαίο στοιχείο εξοπλισμού, επομένω μπορείτε να λάβετε πάρα πολλά διαφορετικά αριθμητικά στοιχεία. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα πρέπει να αναζητήσουμε τα στατιστικά στοιχεία. Τα συλλέγουμε αυτά τα στοιχεία. Αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να κατευθύνουμε τη συζήτηση προς αυτό, να βρούμε αν έχουμε ακριβή στοιχεία και έναν ακριβή μεμονωμένο αριθμό. Ως προς το βάθος, αυτό που σας είπα, ίσως ήταν λίγο βεβιασμένο ή δεν τα είπα καλά. Να το ξαναπώ λοιπόν. Οι διαθέσιμες πληροφορίες από μας, για μας από τον κλάδο και για τα κράτη-μέλη μας λένε ότι στη Βόρεια Θάλασσα το μέσο βάθος επιχειρήσεων είναι 90 μέτρα. Οι γεωτρήσεις γίνονται από αρκετά μέτρα μέχρι περίπου τα 200 στη πλειονότητά τους. Το πιο βαθύ είναι στα 700 μέτρα, αλλά αυτό δεν είναι το πιο χαρακτηριστικό ε, παράδειγμα. Από ό,τι μου λένε, η πλειονότητα γίνεται μεταξύ κάποιων μέτρων και 200 μέτρων και ο μέσος όρος είναι 90 μέτρα. Αλλά υπάρχουν ε, κάποιες ε, μεμονωμένες εξαιρέσεις που φτάνουμε σε βάθη μέχρι τα 700 μέτρα. δεν μπορεί να πάει κάποιος πιο βαθιά, ε, απλώς και μόνο γιατί η Βόρεια Θάλασσα δεν είναι πιο βαθιά. Αν όμως κάποιος βγει πιο έξω, πάει στα νησιά Σέτλαντ κλπ, μπορείτε να πάτε και σε μεγαλύτερο βάθος. Αυτή τη στιγμή βέβαια στην περιοχή αυτή έχουμε μόνο στα Σπάργανα δραστηριότητες και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Μου ζητήσατε κατά πόσο συζητάμε με την Νορβηγία. Έχουμε πολύ στενές επαφές με την Νορβηγία και έχουμε μια συνεδρίαση που σας είπατε των συντονιστών την Παρασκευή και θα συμμετέχουν και οι αρχές της Νορβηγίας, όπως επίσης και οι αρχές εποπτείας των νησιών Φαρόε. Έχουν μια ξεχωριστή αρχή για τα νησιά Φαρόε, η οποία είναι υπεύθυνη μόνο για αυτή την περιοχή. Επίσης με ρωτήσατε τι νομοθεσία ισχύει και πού. Θα πρέπει ίσως να διευκρινίσω και εδώ κάποια πράγματα, διότι και η εθνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία ισχύουν εντός των χωρικών υδάτων, δηλαδή κοντά στις ακτές, η διάκριση που γίνεται και η ακολουθία αυτή που έχουμε στην, ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή στα πρώτα τρία μίλια είναι η πολιτεία υπεύθυνη και τα υπόλοιπα είναι ευθύνη των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Ευρώπη δεν ισχύει αυτό. Η δικαιοδοσία είναι εντό των χωρικών υδάτων. Εκεί ισχύει λοιπόν εθνική νομοθεσία και ε, κατά συνέπεια και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Από εκεί και πέρα μπορεί να έχουμε οικονομικές ζώνες μέχρι τα 200 μίλια εκτός των περιοχών τους και από εκεί και πέρα προεκτείνεται η εγκυρότητα της νομοθεσίας που σημαίνει και πάλι ότι έχουμε προέκτηση όχι μόνο εθνικής αλλά και ευρωπαϊκής νομοθεσίας στις οικονομικές ε, ζώνες ε, μετά από τις οικονομικές ζώνες, συγγνώμη, έχετε διεθνή ύδατα και εκεί έχουμε διεθνή συμβάσεις οι οποίες ισχύουν και έχουν πολύ εκτεταμένες διατάξεις για παραγωγή υδρογονάνθρακα και εξορίξεις. Κάποιες αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιοχές, για παράδειγμα έχουμε τη σύμβαση Όσπαρ για το Βόρειο Ατλαντικό ή έχουν ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και γεωγραφική έκταση. Υπάρχει όμως ένα ρυθμιστικό καθεστώς και για αυτά τα διεθνή Μιλήσατε για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας ε, για τις εξέδρες ε, για να περιμνήσουμε ώστε να έχουμε ίδιες πηγέ πληροφόρηση. Βεβαίω δεν περιμένουμε από την ε, βιομηχανία ή από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Κάνουμε τις δικές μας έρευνες και έχουμε τα δικά μας δεδομένα. Προέρχονται από ανεξάρτητη έρευνα. Δεν έχουμε ακόμη ζητήσει ειδική μελέτη για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών υδάτων, αλλά είναι ένα από τα επόμενα βήματα ε, που σκοπεύουμε να κάνουμε. Ε, τώρα θέλουμε να δούμε τι είδους δεδομένα πρέπει να συλλέξουμε, ποιο είδους πληροφορίες χρειαζόμαστε. Ταυτόχρονα η βιομηχανία και τα κρατη μας δίνουν ε, πληροφορίες και με ξαφνιάζει αυτό που άκουσα ότι ε, ζήτησαν ε, μέλη της Επιτροπής σας στοιχεία από τη βιομηχανία και δεν τα έλαβαν. Ο Επίτροπος έδωσε ένα κατάλογο σημαίνουν προς τους εκπροσώπους των εταιριών του κλάδου στις 11 Μαΐου, σημείων για τα οποία θα θέλαμε περαιτέρω πληροφόρηση. Προσπαθήσαμε να απευθυνθούμε σε όλες τις βασικές πετρελαϊκές εταιρείες στην Ευρώπη, αλλά και στην ε, Ένωση των Παραγωγών Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου και ε, θα απαντήσουν συλλογικά. Δεν ζητούμε απαραίτητα αριθμητικά στοιχεία, αλλά πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση τους, τι εγγυήσει, την πρακτική που ακολουθούν, τη συμπεριφορά τους, την ε, νοοτροπία του ω προς τη διαχείριση κινδύνου. Στις 14 ε, Ιουλίου θα κάνουμε τη δεύτερη συνεδρίαση μαζί τους, ε, όπου θα έχουμε συλλογικά τι απαντήσει του κλάδου. Και ε, αυτό που θα φροντίσουμε είναι να επικρατήσει η διαφάνεια σε σχέση με αυτά που κάνει ε, η βιομηχανία. Όχι να μας καθησυχάσουν μόνο και να επαναλάβουν την ε, δέσμευσή τους. Όχι βέβαια ότι δεν είναι και σημαντική η δέσμευση της βιομηχανίας, αλλά πέραν αυτού πρέπει να συζητήσουμε τα βήματα που κάνουν ε, μετά την ε, καταστροφή, ούτως ώστε να ενισχύσουν ε, την ασφάλεια των επιχειρήσεών τους και τη διαφάνεια. Πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό αναμφισβήτητα η βιομηχανία κάνει κάποια βήματα, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει και προβολή αυτών των ε, βήματων για να τα μάθει και το ευρύ κοινό και όλοι οι ενεχόμενοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν στη συνέχεια και εύστοχα ερωτήματα, αν χρειαστεί. Αυτό θα ενισχύσει και τη συμμόρφωση προς την ομοθεσία. Είναι ένα από τα σημεία που έχουμε στενή συνεργασία με τη βιομηχανία παρομοίως με τις εθνικές αρχές ε, θέλουμε να δούμε πώς επισταμένα ε, κάνουν την παρακολούθηση και την ε, εποπτεία της διαδικασίας. Συμφωνούμε με την προσέγγιση τους Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επέμβει μόνο όταν μπορεί να προσθέσει κάτι, να έχει προστιθέμενη αξία σε σχέση με τις προϊούσες ε, διαδικασίες, δηλαδή να προσθέσουμε άλλο ένα στρώμα ε, ασφάλειας, διαφάνειας ή συμμόρφωσης ε, προς την νομοθεσία. Αυτή είναι η γενικότερη προσέγγισή μας. Uh, ε, αναφερθήκατε σε μια πιθανή απαγόρευση των επιχειρήσεων ε, και τη σύσταση ταμείου και ε, την αλλακτική πρακτική υποχρεωτικής εγκυοδοσίας. Μάλιστα, ναι, όλα αυτά είναι πιθανά μέτρα Δεν νομίζω όμως ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο για να αποφανθούμε, δηλαδή να τοποθετηθούμε σχετικά με το ποιο είναι το καταλληλότερο κατά τη γνώμη μας μέτρο. Είναι σημαντικό να δούμε ποια μαθήματα ε, ε, έχουν, ε, ποια διδάγματα έχουν αντλήσει τα κράτη-μέλη από το ατύχημα, ποιες είναι οι δεσμεύσεις της βιομηχανίας και αν εξακολουθούν ευθύς να υπάρχουν κενά και μπορούμε να αναλάβουμε δράση σε νοσιακό επίπεδο, ναι, ναι, είμαστε φιλόδοξοι και να το πράξουμε. Είμαι σίγουρος ότι δεν κάλυψα όλες τις ερωτήσεις, προσπάθησα όμως. Θα καλύψω το, τα περισσότερα από τα σημεία που έγιραν ε, οι συνάδελφοι. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Εφόσον ε, εκτελώ χρέη Προέδρου, θα μου επιτρέψω κι άλλη μια ερώτηση. Ε, πώς ακριβώς συνεργάζεστε με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Περιβάλλοντος. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Και σε πολιτικό επίπεδο και σε ενδοϊπηρεσιακό επίπεδο. Σε 11 Μαΐου, σε αυτή τη συνεδρία που σας έλεγα, ο πρόεδρος Έτιγκερ αρμόδιος για την ενέργεια και η Επίτροπος Γεωργίευα που ασχολείται με την πολιτική προστασία ε, συμμετείχαν. Ο Επίτροπος Ποτόσνικ δεν ήταν στις Βρυξέλλες τότε, αλλά ο επικεφαλής ε, του επιτελείου του επίσης ήταν στη συνεδρίαση. Ε, δηλαδή συμμετείχε η πολιτική ηγεσία εξ αρχής και για τα επόμενα βήματα υπάρχει στενή συνεργασία σε ενδοϊπηρεσιακό επίπεδο. Η αναθεώρηση της νομοθεσίας ε, που τώρα ε, διεξάγεται από διάφορες υπηρεσίες. Ε, λοιπόν, υπάρχει στενή συνεργασία συγκεκριμένα με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ περιβάλλοντος. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λάβαμε και επιπρόσθετες παρατηρήσεις από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Υπάρχει έντονη συνεργασία. Σας είπα ότι προτιθέμεθα να δημιουργήσουμε και μια ενδοϊπηρεσιακή ομάδα όπου θα εκπροσωπηθούν όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες και φυσικά και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και μπορώ να διαβιβάσω Ενδεχομένω και τις ανησυχία σα ότι κρύβεται πίσω μας ε, η γαμαδέλτα περιβάλλοντο, ότι αποφεύγει τα φώτα της ε, δημοσιοτητα Δεν ισχύει αυτό, σα διαβεβαιώ. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώνουμε έτσι αυτό το σημείο. Επεννούμε στο τελευταίο σημείο για σήμερα. Προφορική ερώτηση 2010 06 των Chris Davis και Κορίν Λεπάζ σχετικά με την οδηγία για, τα, ε, για την ποιότητα των καυσίμων για τα εφαρμοστικά μέτρα άρθρο 7α ασφαλτούχος άμμος. Έχουμε εκπρόσωπο από τη Γενική Διεύθυνση ε, Κλιματικών Αλλαγών. Είναι ο, ο τμηματάρχης Φίλιπ Όουεν συγκεκριμένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους που μα δίνετε την δυνατότητα να έρθουμε εδώ σήμερα και να σας ε, παρουσιάσουμε τι συζητιζόμενη εργασία εφαρμογή <clears throat> μέσα στα πλαίσια και με την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων. Όπως ξέρετε, μία από τις ε, προϋποθέσεις της ε, ε, οδηγίας είναι να υπάρχει μια μεθοδολογία για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Υπάρχουν εργασίες που συνεχίζονται και είναι σαφές ότι η μεθοδολογία που προετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή <clears throat> έχει μια απόλυτη ισορροπία μεταξύ της, ε, του πολύπλοκου διοικητικού της χαρακτήρα και της αποτελεσματικότητά της. Έχουμε εργαστεί εδώ και αρκετό καιρό για τη μεθοδολογία. Πέρσι το καλοκαίρι αρχίσαμε τη διαδικασία διαβούλευση ε, μέχρι και το φθινόπωρο. Το Γενάρη φέτος είχαμε μια συνεργασία με τους ενδιαφερόμενου στα κράτη-μέλη και τον Μάρτι συζητήσαμε και ένα έγγραφο των κρατών μελών πριν καταλήξουμε στις συμπεράσματα. Ο στόχος της Κομισιόν είναι αυτή η μεθοδολογία να υιοθετηθεί μέσα τα όρια του 2010 και ξέρω ότι είχατε ήδη τη δυνατότητα να ε, συζητήσετε το θέμα αυτό με την Επίτροπο Χέντεγκάρκ την περισμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Τούτου λεχθένως θα ήθελα να αναφερθώ στα συγκεκριμένα θέματα της ερώτησης. Πρώτον, στο διαβουλευτικό μας έγγραφο πέρσι συμπεριλάβαμε με κάποιες αξίες όσον αφορά τις ε, ασφαλτούχους άμμος. Η Κομισιόν ίδια δεν έκανε όμως ε, μια αξιολόγηση των ε, καυσίμων που παράγονται από ασφαλτούχους άμμος, μια που αυτό είναι κάτι που αφορά το Κοινό Κέντρο Ερευνών και για το οποίο έχουν ε, οριστεί αξίες ποιότητας μέσα στα πλήσια του εγγράφου που είχα προναφέρει. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένες ε, εκθέσεις από διάφορες ομάδες που ορίζουν κάθε μια την αξία που θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει και θα πρέπει να εξετάσουμε εις βάθος αυτές τις αξίες. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε την κατάλληλη μεθοδολογία ακόμα. Δεν έχουμε τελειοποιήσει τίποτα και γι' αυτό δεν έχουμε φτάσει σε συμπεράσματα όσον αφορά ποια θα είναι η μορφή που θα έχει η πρόταση. Συνεπώς σήμερα δεν μπορώ να σας δώσω την τελική εκτίμηση. Ε, Ιδίω όσον αφορά τις ασφαλτούς άμμους. Μπορώ να σας πω όμως η Κομισιόν θα αναλύσει όλες τις εναλλακτικέ και θα σας υποβάλει τη σωστή πρόταση. Οπωσδήποτε θεωρούμε ότι ο στόχος του 6% θα καλυφθεί με την χρήση αηφόρων μορφών ενέργειας και ε, ανανοσίμων πηγών ενέργειας. Εάν τελικά υπάρξει σημαντική ε, αύξηση εισαγωγών ασφαλτούχων άμμων και δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι αυτή τη στιγμή αλλά εάν γινόταν λέω θα σημαίνει ότι θα πρέπει να δράσουμε περισσότερο και να αντιδράσουμε με μεγαλύτερη χρήση βιοκαυσίμων για να πετύχουμε τους στόχους που έχουν οριστεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, e, Ευχαριστώ. Θα έχουν τον Κρίς Τέιβις πρώτος και μετά ο κύριος Κρέτον και τρίτος ο κύριος Εκχάουτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μα είπε η Κομισιόν δηλαδή ότι δεν μπορεί να απαντήσει και ότι δεν έχουν ολοκληρώσει τη μελέτη. Δεν είναι πολύ κατάλληλη αυτή η απάντηση, αλλά την καλωσορίζω γιατί μας δείχνει ότι ακόμα είναι ανοιχτή η διαδικασία για επιδράσεις. Ε, Μελετέται προσεκτικά και δεν έχουν ληφθεί ακόμα αποφάσεις. Ίσως η συνάντηση με τον Επίτροπο Ελευθερών Εβδομάδα ήταν χρήσιμη. Βέβαια ξέρει η Κομισιόν ότι υπήρχαν διάφορες εικασίες που ακούστηκαν ότι υπάρχει επίδραση από λόμπι, από την καναδική κυβέρνηση, από τη ΣΕΛ για να μειωθούν οι στόχοι που έχουν αρχικά προταθεί στο πρώτο έγγραφο. Έγινε μία αναφορά στην αξία που προτάθη στο έγγραφο αυτό ότι προήλθε από κάποια συγκεκριμένη πηγή. Εγώ έχω σημειώσει εδώ ότι λέγεται ότι έχουν γίνει πάνω από 12 μελέτε από την κρατική κυβέρνηση και την ΣΕΛ και οι περισσότερες από τις μελέτε αυτές έβαλαν μια αξία 160 106 συγγνώμη, γραμμαρίων για τους ασφαλτούχους άμμους. Η Κομισιόν προτείνει 107. Ε, εκεί στα όρια βρίσκεται. Αλλά προφανώς δεν έχουμε καμία συγκεκριμένη απάντηση της Κομισιόν αυτή τη στιγμή για το θέμα. Το ουσιαστικό θέμα είναι σαφές. Ο στόχος της νομοθεσίας είναι να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Και αν μπορούμε να έχουμε παραγωγή ακαθαριστείου πετρελαίου από, από τις ασφαλτούχους άμμους αυτή, ε, δεν νομίζω ότι πετυχαίνουμε το στόχο. Ελπίζω να συνεχίσει η Κομισιόν να εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή. Κατανοείται ότι υπάρχει έντονη πολιτική άποψη εδώ στην Επιτροπή μας και σε όλο το Κοινοβούλιο ότι αν η Κομισιόν υποβάλει κάποια ε, πρόταση επιτροπολογία που δεν λαμβάνει υπόψη τις δικές μας ανησυχίε, ο κίνδυνος είναι όλη η νομοθεσία να απορριφθεί. Χαίρομαι που ο Επίτροπος προφανώς το μελετάει το θέμα προσεκτικά και περιμένω να δω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τις ερωτήσεις και τα σχόλια του Chris Davis. Για να πάω λίγο περαιτέρα, διότι μου φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι βέβαιοι για τα στοιχεία και το ίδιο είχαμε και στα βιοκαύσιμα. Γι' αυτό και το, στα βιοκαύσιμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε μια υβριδική προσέγγιση και εκεί μπορούμε να επιλέξουμε μια υψηλή τιμή και να έρθουν οι επιχειρήσεις και να αποδείξουν ότι η δική τους παραγωγή σχετίζεται με χαμηλότερη τιμή. Και έτσι έχουμε και πολλά στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ανάλογη τεχνογνωσία γιατί έχει ξαναχρησιμοποιηθεί στο παρελθόν λοιπόν αυτή η προσέγγιση. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν στις συζητήσεις που κάνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο συζητάτε μια τέτοια υβριδική προσέγγιση. Και επειδή ε, εξετάζετε τη δυνατότητα ενός συντελεστή για την ασφαλτούχο άμα, κατά πόσο θα λάβετε υπόψη σας και τη ε, ε, χρήση της γης. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι στον Καναδά έχουμε μεγάλη χρήση εκτάσεων και αυτό φυσικά ε, έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα και φυσικά έχουμε και τη Μαδαγασκάρη και άλλες περιοχές που είναι πολύ σημαντικές για τη βιοπικιλότητα. Ευχαριστώ. Κύριος Eichhout. Uh, Ευχαριστώ τον Φίλιπ Όουεν για τις ε, απαντήσεις του. Δυστυχώ δεν ήσασταν σε θέση να μα δώσετε όλε τι απαντήσεις που μας είπατε και αυτό απάντηση είναι. τέλο πάντων. Επανέρχομαι σε κάτι που είπατε. Είναι να βρείτε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ακρίβεια και την σωστό καταμερισμό του διοικητικού άχθους. Ωραία, αν το θέτετε έτσι, όλοι επιθυμούμε αυτή την ισορροπία. Αλλά δεν κατανοώ πώ επιχειρηματολογείτε ε, το διοικητικό άχθο. Υπάρχουν πολλές μελέτες ε, που σαφώς ε, καταδεικνύουν το συντελεστή για τι εκπομπέ. Οπότε ε, το να έχουμε μία αυτόματη τιμή ε, σε ολόκληρο τον πίνακα που έχετε με τις τιμές ε, για το αργό πετρέλαιο, για τα υγρά καύσιμα, για το φυσικό αέριο που μετατρέπει σε υγρό καύσιμο. Άντε να βάλουμε και άλλη μία τιμή εκεί δεν νομίζω ότι είναι και τόσο βαρύ διοικητικό πώ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί για τι εταιρείε των ε, καυσίμων, των ορυκτών καυσίμων. Αλλά έχουμε και την οδηγία για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Έχουμε ολόκληρα παραρτήματα για τι ε, ε, κανονικέ τιμέ, για τι ενεργειακέ πηγέ. Μία φοβερή σειροή Καλό είναι να ορίσουμε μια αξία, γιατί ξέρουμε ότι και η βιομηχανία ορεικτών καυσίμων πρέπει να εξετάσει πολλά παρατήματα για να καταλάβει ποιε είναι οι σωστέ τιμέ. Ωραία, μπορεί η βιομηχανία να μα λέει ότι δεν ξέρουν ποιε είναι οι εκπομπέ τη ασφαλτούχου άμμου. Ε, συγγνώμη, αλλά ε, από τα διηληστήριά τους ξέρουν ακριβώς ποιες είναι οι εκπομπές γιατί το πληρώνουν. Τα έχουν ήδη τα έγγραφα, πόσο έχουν πληρώσει τους ισολογισμούς τους, δηλαδή πόσο έχουν πληρώσει στα διηληστήρια, οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να αναγνωρίζουν το συντελεστή για τις εκπομπές. Ε, ωραία, να τη βρούμε την ισορροπία, αλλά δεν βρίσκω ότι συνιστά αυτό μεγάλο διοικητικό άχθος ούτε για τις εταιρείε. Και μας λέει ο κύριος Όβεν ότι ε, προς το παρόν είναι μικρή εισαγωγή της άμμου αυτή. Ναι, αλλά για δείτε τα αποθέματα της ΣΕΛ, το 25% είναι ασφαλτούχος άμμος. Το 1 τέταρτο. Οπότε στο μέλλον αυτόματα ε, θα ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο καυσίμων που χρησιμοποιούμε για τα οχήματά μας. Χρειάζεται να ορίσετε ε, τιμή. Είναι εύκολο, έχουν γίνει οι μελέτες, εύκολο μπορούν να το λάβουν υπόψη και οι εταιρείες. Οπότε καλωσορίζω αυτό το βήμα που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά περιμένω σε λίγες εβδομάδες ε, να έχουμε ένα νέο πίνακα που θα έχει προσθεθεί η τιμή για την ασφαλτούχο άμμο. Όλοι θέλουμε μειώσεις. Ε, αυτός είναι εξάλλου ο πρωταρχικός στόχος της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων, έτσι. Ευχαριστούμε. Η Λίντα Μακέβαν. Ο συνάδελφος με πρόλαβε, είπε πολλά, οπότε θα πω μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, πριν από τις συνεδρίες που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ακούγαμε ότι δεν γίνεται να κάνουμε τίποτα για την ασφαλτούχο άμμο. Και τώρα μας λέει ότι είναι ανοιχτό το ζήτημα, εκκρεμεί και ακόμη το επεξεργάζονται. Ωραία, συνιστά αυτό πρόοδο, συμφωνώ. Αλλά ε, καλή εξήγηση δεν είχαμε γιατί εξαφανίστηκε ξαφνικά το αρχικό στοιχείο από πέρσι. Δεν θέλουμε να περάσουμε λάθος πολιτικό μήνυμα ε, ότι θέλουμε η ασφαλτούχος άμμος ε, να γίνει βασική πηγή πετρελαίου. Αν είστε σοβαροί για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών πρέπει να το ρυθμίσουμε το ζήτημα. Εμεί θα μείνουμε αμετακίνητε στη θέση μα. Είναι σοβαρό το, το ζήτημα, το πιστεύουν όλε οι πολιτικέ ομάδε και περιμένουμε νέα σα επιτροπή. Ο Φίλιπ Όουεν θα ήθελε να δευτερολογήσει. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Από τα σχόλια των συναδέλφων ε, θα ξεχωρίσω δύο ερωτήματα και θα απαντήσω. Λοιπόν, τα βιοκαύσιμα και προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, αυτό ήταν το έγγραφο διαβούλευσης, αλλά τελικά δεν έτυχε ευρεία ε, αποδοχής, γι' αυτό και δεν ακολουθήσαμε τις προτάσεις. Τα κράτη-μέλη και οι εμπλεκόμενοι εταιροί ήθελαν μια αυτόματη τιμή, default value, γιατί είναι πιο εύκολα εφαρμόσιμη. Για τον Καναδά και τα Ε, και τα εγκυοβελτιωτικά ε, έργα ε, για μένα εκρεμεί το ζήτημα και το έχω συζητήσει επανειλημμένα με τους Καναδούς εταίρους, αλλά δεν έχουμε άλλα νέα. Για αυτό το θέμα της προσέγγισης της αυτόματης τιμής, ναι, ένας από τους στόχους να μειώσουμε το διοικητικό βάρος. Γιατί οι προμηθευτές καυσίμων που πρέπει να αναλάβουν και την ευθύνη θα έχουν να κάνουν με ένα μόνο αριθμητικό στοιχείο, με μία τιμή και όχι να παρακολουθούν όλη την αλυσίδα για να ε, προσδιορίσουν ποια στάδια μετατροπής έχει υποστεί το καύσιμο και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό προτιμούμε τον, ε, την αυτόματη τιμή και θεωρούμε ότι συνεπάγεται μικρότερο διοικητικό άχθος Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλο απόθεμα ασφαλτούχου ε, ε, άμμου ε, στον Καναδά. Πρέπει να δούμε τις εμπορικές δροές, πώς θα μετεξελιχθούν. Αλλά βάσει των πληροφοριών που έχουμε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, δεν υπάρχουν ακόμα εισαγωγές στην Ευρώπη. ανεπεξέργαστης ασφαλτούχου άμμου. Ευχαριστούμε. Ε, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση. Στις 13 Ιουλίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 θα διεξαχθεί η επόμενη συνεδρίασή μας και επίσης στις 14